Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ, καλημέρα. Και να έχετε τις κάρτες σας, γιατί θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Χθες δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις ψηφοφορίες, οπότε συνεχίζουμε το σημείο 12, κοινό σύστημα για την εγγραφή των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών. Αρχίζουμε την πληροφορία Τροπολογία 14, 17, 18 και 16. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε την 27. Ε, θε, όπως σαλφος συνάδελφος Κλάς. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 12-4. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34. Α, έχει απορριφθεί. Έχει απορριφθεί το πρόβλημα. 34 υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Α, ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 34 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 9 υπέρ 16 κατά. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 και 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46, 47 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Το άκουσα, το άκουσα Καρλ Ωραία, ας ελέγξουμε την 47. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρία και 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 41 με την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 κατά τμήματα το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα Α, δεν θα ψηφιστεί. Γιατί ενεκρίθησαν οι προηγούμενες δύο. Τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 με προφορική τροπολόγηση υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται με την προφορική τροποποίησή της. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε, ασαφές. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ε, 51. Όχι, 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 62 Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65, 66, 67 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 12 υπέρ. 12 κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 20 παρακαλώ ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Καλά, ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 24. Νομίζω ήταν ε, ο ίδιος συσχετισμός. Αλλά προς την άλλη κατεύθυνση. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ελέγξαμε την 24 και ενεκρίθη. Οπότε 25 καταπίπτει. 19 με την προφορική τροποποίησή της. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 19 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Ωραία. Τώρα να κάνουμε την τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Συγχαρητήρια ε, στον εισηγητή 35 στην εισηγήτρια. 35 ε, υπέρ, 3 κατά. Οπότε κλείσαμε. Και περνάμε στο άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπου θα χρειαστούμε αρκετό χρόνο γιατί έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες. Παρακαλώ μείνετε, ε, ευχαρίστως. Αλλά Ας περιμένουμε λίγο. Ωραία, νομίζω ησύχασαν τα πράγματα. Θα πρότεινα λοιπόν τώρα να έχουμε τη συζήτηση για το γκάπνο. Και πρώτος, Πρώτη η εισηγήτρια. Λίντα, είσαι έτοιμη. Λίντα Μακάρδον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι γαλινεύουν οι συνάδελφοι και μπορώ να λάβω το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι. Τα άσχημα νέα πρώτα πάνω από 1.300 τροπολογίες έχουμε μόνο από τη δική μας Επιτροπή για την Οδηγία για τα καπνικά προϊόντα. Τα καλά νέα είναι ότι πολλές τροπολογίες είναι ταυτόσιμες και πολλές από αυτές αφορούν τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Δεν θα σταθώ στα θέματα αυτά γιατί νομίζω πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την πρόταση της Κομισιόν. Είναι πολλά θέματα όπου πρέπει να επανέλθουμε στη διαδικασία συναπόφασης όπως ζητούν οι συνάδελφοι. Είναι όλα αυτά τα θέματα λοιπόν για τις ε, κατεξουσιοδότηση αλλά πρέπει να τις προσέξουμε για να μην θυγούν οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Ίσως ε, μπορείτε να κάνετε τα πηγαδάκια σας έξω και να αφήσετε την εισηγήτρια να παρουσιάσει την έκθεσή της και να μας δώσει και τις απόψεις της για τις τροπολογίες μέσα σε ένα πιο γαλήνιο κλίμα. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα και πρέπει να έχει την κατάλληλη προσοχή, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, λέει και η Λίντα. Έχουμε πολλέ τροπολογίε, όπως σας είπα. Δεν πηγαίνουν όλες προς την διακατεύθυνση οι τροπολογίες για πολλά από τα κέρια θέματα, αλλά υπάρχουν κάποιες κοινέ κατευθύνσεις για πολλές τροπολογίες είναι κάποιοι συνάδελφοι, λίγοι, οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά να ακυρώσουν όλη την πρόταση της Κομισιόν μέσω τροπολογιών. Να τη διαγράψουν, να διαγράψουν τα άρθρα της πρόταση της Κομισιόν. Αλλά οι περισσότεροι δέχονται το κύριο επιχείρημα της Κομισιόν που λέει ότι πρέπει να δράσουμε και πρέπει να θυμηθούμε γιατί αναλαμβάνουμε θράση. Αυτοί που νομίζουν πρέπει να ακυρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία της Κομισιόν, ξέρετε ότι όλα τα κράτη-μέλη μας έχουν προσυπογράψει την οδηγία πλαίσιο για την, την σύμβαση πλαίσιο για τον έλεγχο των καπνικών προϊόντων που ζητά από τα κατημέλη να αναλάβουν δράση. Και όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας συνεδρίαση, μπορεί να θεωρούμε ότι προηγούμεθα έναντι του υπόλοιπου κόσμου σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση, τα ρυθμιστικά θέματα, για τον καπνό δεν έχουμε προχωρήσει. 28% είναι το ποσοστό των καπνιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι γύρω στα 20%, 17,5% στον Καναδά. Δεν είμαστε λοιπόν μαζί με τις αναπτυγμένες χώρες σε ό,τι αφορά τη μείωση του πληθυσμού των καπνιστών. Φυσικά μειώνεται αυτό το ποσοστό, αλλά όχι αρκετά γρήγορα και δεν μειώνεται με τον ίδιο ρυθμό όπως στις Πολιτείες, στη Βραζιλία, τον Καναδά και πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής που κάνουν τώρα πολύ σημαντικά βήματα για να αντιμετωπίσουν το θέμα του καπνίσματος. Και υπάρχουν και ανησυχητικές ε, τάση σε ορισμένε χώρε όπου μειώνεται μεν το γενικό ποσοστό των καπνιστών στον πληθυσμό, αλλά αυξάνεται για του νέου. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε αυτή την νομοθεσία, να κάνουμε λιγότερο ελκυστικά τα καπνικά προϊόντα για του νέου, να μην δημιουργηθεί μια νέα γενιά καπνιστών από του νέου, αυτό είναι ο στόχο μα, και 99% των ε, φεριακλείδων καπνιστών που δεν, θέλουν να, δεν μπορούν να σταματήσουν το κάπνισμα, δεν θα θέλαν τα παιδιά του να γίνουν και αυτοί οι καπνιστές. Έχουμε μια ευθύνη λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτή την αύξηση των καπνιστών μεταξύ των νέων. Πολλές τροπολογίες λοιπόν έχουμε. Θα εστιάσω στους τομείς όπου βρίσκονται οι περισσότερες τροπολογίες και όπου μπορεί να θέλουν να σχολιάσουν οι συνάδελφοι και θέλω να ακούσω και τις απόψεις αυτών που έχουν καταθέσει τροπολογίες για να τις εξηγήσουν καλύτερα ενώπιον της Επιτροπής μας. Κάποιες από αυτές τις τροπολογίες δεν έχουν αιτιολόγηση επαρκή. Το θέμα των συστατικών τι μπορεί να βάλει κανείς σε ένα τσιγάρο. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Μέχρι τώρα όλα αυτά ήταν κάπως αδιαφανή. Ο κ. Φλόρενς έχει εργαστεί για πολλά χρόνια σε αυτό το θέμα να καταλάβει τι περιέχουν τα τσιγάρα. Είναι απαραίτητο να ξέρουν οι δημοσίες αρχές τι περιέχουν ακριβώς τα τσιγάρα. Έχουμε τροπολογίες που ξεκινούν από τους συναδέλφους που θέλουν να βελτιώσουν την ε, <clears throat> υποβολή αναφορών από τα κράτη-μέλη Προβλέπετε ότι οι κυβερνήσει πρέπει να, να παίρνουν στοιχεία από τι εταιρείε και να τα διαβάζουν στην Κομισιόν, η οποία θα τα αναλύει και θα βλέπει αν χρειάζεται περαιτέρω δράση. Κάποιοι συναδέλφοι έχουν ε, κάνει μια πρόταση για ένα θετικό κατάλογο συστατικών. Δηλαδή να μπορεί κανεί να βάλει στα τσιγάρα μόνο τι ουσίε που βρισκόνται στο θετικό κατάλογο. Και θα ήθελα να ξέρω η Κομισιόν γιατί δεν έχει προτείνει κάτι τέτοιο και πώς αντιδρούν στους συναδέλφους οι οποίοι έχουν προτείνει το θετικό κατάλογο. Δεν είμαι εναντίον τη ιδέα. Αυτή θέλω να δω όμως πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ένα άλλο σημαντικό αμφιλεγόμενο θέμα, το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, είναι το θέμα των ουσιών που προσθέτουν γεύση στα τσιγάρα, πέρα από τα άλλα συστατικά. Η, Κομισιόν δεν εμποδίζει, η πρόταση της Κομισιόν δεν εμποδίζει να προστίθεται ζάχαρη στα καπνικά προϊόντα γιατί αυτό μπορεί να γίνει για τα καπνά τα οποία καλλιεργούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι συνάδελφοι με τροπολογίε ζήτησαν να απαγορευτούν όλα αυτά τα πρόσθετα γλυκαντικά, οτιδήποτε κάνει πιο εύγευστα τα τσιγάρα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουμε στην πρόταση της Κομισιόν. Κατανοώ αυτό που λένε οι συνάδελφοι ότι δεν πρέπει να γίνουν ιδιαίτερα εύγευστα τα τσιγάρα, αλλά ήδη ουσιαστικά εισάγουμε καπνά τα οποία έχουν προσθήκη ζάχαρης και δεν μπορούμε να το σταματήσουμε σε, πρέπει να το σταματήσουμε σε αυτό το επίπεδο και όχι στο τελικό καταναλωτή. Τα βελτιωτικά γεύσεις. Οι περισσότεροι δέχονται την γενική απαγόρευση γεύση σοκολάτα, φράουλα κτλ. Αυτά είναι μικρέ αγορέ προ το παρόν. Δεν θέλουμε φυσικά αυτή η αγορά να διευρυνθεί. Αλλά ορισμένοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν και στη Μενθόλη είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια εξαίρεση για τη μενθόλη σε σχέση με τις άλλες βελτιωτικές ουσίες. Να σας υπενθυμίσω ότι εγώ νομίζω και η μενθόλη θα πρέπει να απογορευτεί γιατί η Επιστημονική Επιτροπή με μια έκθεση 100 σελίδων το 2010 κατέδειξε ότι η μενθόλη έχει χαρακτήρα ελαφρού αναισθητικού εμποτίζει το βήχα και επιτρέπει βαθύτερη εισπνοή. Η FDA, η Food and Drug Administration των Πολιτειών, θεωρεί ότι η μεθόλη μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο πειραματισμό με τα τσιγάρα και να ευνοήσει το κάπνισμα και ότι απευθύνονται ιδιαίτερα στους νέους. Γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει κανείς με τσιγάρα που έχουν μενθόλη όταν ξεκινάει κανείς το κάπνισμα. Έχονται λοιπόν τις τροπολογίες που έχουν πει πολλοί συνάδελφοι τη θέση τους. Αλλά είναι γεγονός ότι τα τσιγάρα με μενθόλη έχουν διευρυνόμενη αγορά γιατί προσελκύουν τους νέους. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που δεν θέλουμε. Να είναι περισσότεροι οι νέοι οι οποίοι καπνίζουν λόγω των σιγάρων, σιγαρέτων με μενθόλη. Η Γερμανία και η... το Βέλγιο έχουν απαγορεύσει ήδη τη μενθόλη. Η Βρασιλία κάθε μορφή βελτιωτικών της γεύσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κάνουν μια γενική απαγόρευση, αλλά τα λόμπι οδήγησαν στην ε, εξαίρεση της μενθόλης ως βελτιωτικού γεύσης. Και άλλες χώρες τώρα διαμφισβητούν αυτά τα οποία έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες με το επιχείρημα ότι είναι διάκριση εναντίον των άλλων ε, τσιγάρων με βελτιωτικά γεύση, όπως τον Ινδονησιακό Κρέτεκ, παραδείγματο χάρη. Εάν λοιπόν κάνουμε μονάχα μια εξαίρεση για την μενθόλη, τότε είμαστε ανοιχτοί σε διαφυσβήτηση από άλλους οι οποίοι θα πούν γιατί όχι εξαίρεση και για αυτά που έχουν ε, σοκολάτα ή φράουλα ή κάτι άλλο. Είναι γενικό λοιπόν το θέμα αυτό της ε, ε γεύσης και έχουμε και τα θέματα για το σνούς. Το σνούς αυτή τη στιγμή επιτρέπεται μόνο στη Σουηδία και νομίζω και στην Φιλανδία. Μπορεί να μου το διευκρινίσει η Κομισιόν. Αλλά είναι ένα σουηδικό θέμα ουσιαστικά. Σουηδία έχει μια εξαίρεση από τις ευρωπαϊκές συνθήκες και έχει το δικαίωμα να πουλάει σε εσωτερικό επίπεδο το σνούς. Κάποιοι θέλουν να επιτρέψουν το σνούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ δεν το υποστηρίζω καθόλου, άλλοι συνάδελφοι λένε εντάξει, άμα είναι μονάχα ένα σουηδικό θέμα, τότε θα πρέπει να υπάρχει ρύθμιση του σνούς μόνο στη Σουηδία. Και υπάρχουν κάποιε τροπολογίε για το θέμα αυτό, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Έρχομαι τώρα στη συσκευασία και τις ετικέτες. Εδώ υπάρχουν πολλές τροπολογίες. Πολλοί πιστεύουν ότι η Κομισιόν προχωρά υπερβολικά, επιβάλλει ιδιαίτερα για το πώς πρέπει να είναι οι προειδοποιήσεις, πώς πρέπει να είναι η συσκευασία, τι μορφή πρέπει να έχουν όλες αυτές οι έγγραφες προειδοποίησεις. Κατανοώ αυτές τις τροπολογίες που λένε παραγωγή χάρη. Το είπαν κάποιοι Πορτογάλοι συνάδελφοι που τα πακέτα τους είναι κάπως μικρότερα από τα άλλα πακέτα δεν πρέπει να μας τρελάνει τώρα το αν είναι ακριβώς το ίδιο μέγεθος ή όχι η προειδοποίηση σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν τροπολογίες από πολλούς συναδέλφους επίσης για τον καπνό που το στρίβει κανείς μόνος του. Λέει η Κομισιόν πρέπει να είναι μονάχα, να πουλιέται μονάχα σε σακουλάκια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον καπνό που είναι σε κουτιά, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι μόνο σε σακουλάκια και όχι σε κουτιά. Επομένω πρέπει να μπορούμε να δεχτούμε και αυτή τη δυνατότητα να υπάρχουν και κυλινδρικά κουτιά με καπνό που στρίβει κανεί μόνο του. Πρέπει επίση να σκεφτούμε ιδιαίτερα μέχρι ότου μειώσουμε το μέγεθος, την επιφάνεια που καλύπτουν οι φωτογραφίες και οι προειδοποίησεις. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο λόμπι εναντίον αυτών. Γιατί ξέρουν οι τσιγαροβιομηχανίες ότι είναι αποτελεσματικές αυτές οι φωτογραφίες. Υπάρχουν 9 ή 10 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρησιμοποιούν φωτογραφίες στη συσκευασία και 63 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο το κάνουν. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινοφανές. Και δεν θα δεχτώ αυτή την ιδέα που λένε ορισμένοι ότι αυτό είναι ένα καινούριο, κάτι το καινούριο να βάζουμε φωτογραφίε. Το Συμβούλιο δεν θα το δεχτεί γιατί είναι κάτι που χρησιμοποιείται από πάρα πολλέ χώρε σε παγκόσμιο επίπεδο και άλλε χώρε θα το εισαγάγουν τώρα αλλά είναι και το θέμα του μεγέθους. Δεν έχω ένα πακέτο τσιγάρων μαζί μου, αλλά μερικά από τα πάρα πολύ ε, μικρά και λεπτά πακέτα έχουν φωτογραφίες τόσο μικρές που δεν μπορεί κανείς να τις δει καλά καλά. Όλα τα στοιχεία και είδα τις τροπολογίες από κάποιους συναδέλφους που λένε ότι δεν έχουν καμιά επίδραση φωτογραφίες. Ίσα ίσα έχουμε πολλά στοιχεία ότι οι φωτογραφίες είναι αποτελεσματικές. Γι' αυτό πολλέ από τι κυβερνήσει έχουν εισαγάγει τι φωτογραφίε και άλλε κυβερνήσει θέλουν να προσθέσουν τι φωτογραφίε όταν εγκριθεί αυτό το νομοθέτημα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να παραμείνουμε με τι φωτογραφίε και να κρατήσουμε το μέγεθο των προειδοποίησεων. Υπάρχουν πολλέ πιέσει για τι προειδοποίησει. Αν λένε τα λόμπι ότι, όπω λένε οι τροπολογίες ότι δεν έχει σημασία το μέγεθο των προειδοποίησεων, γιατί θέλουν να μειώσουν το μέγεθος αυτό, άμα δεν του μοιάζει. Για τη συσκευασία έχουμε πάλι τροπολογίε που θέλουν να διαγράψουν όλη την πρόταση της Κομισιόν και τροπολογίε που περνάνε πιο μακριά από την πρόταση της Κομισιόν. Παραδείγματο χάρη να υπάρχει ε, μια ομοιόμορφη καινή συσκευασία χωρίς ε, φωτογραφίες και διαφημίσεις όπως στην Αυστραλία. Άλλοι θέλουν να καταργηθεί η διάκριση μεταξύ τσιγάρων που στρίβει κανείς μόνος του και των άλλων προϊόντων. Θέλουν όλα τα προϊόντα να έχουν ακριβώς την ίδια ετικετοθεσία και να μην αναφέρεται η διαφοροποίηση αυτή. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Επίσης, το θέμα των την απλή συσκευασία, τη συσκευασία χωρίς ενδείξεις και διαφημίσεις. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Και αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η χνηλασιμότητα, στοιχεία ασφαλείας. Οι περισσότεροι συνάδελφοι κατανοούν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να δεχτώ όμως ότι με τις μεγάλες προειδοποίησεις, μεγάλου σχήματος προειδοποίησης, αυτό αυξάνει την ε, παραποίηση των ε, κουτιών τσιγάρου. Νομίζω ότι η Κομισιόν θα έρθει αυτή τη βδομάδα με μια πρωτοβουλία και ίσως μπορεί να μας το εξηγήσει τώρα για να αντιμετωπιστεί η παραποίηση και τα λαθρέα τσιγάρα. Και έχουμε εδώ πέρα και μια ολόκληρη παράγραφο για να κάνουμε πιο εύκολη την ειχναλασιμότητα των τσιγάρων και να έχουμε περισσότερα στοιχεία ασφάλειας. Διαμεθοριακές πωλήσει. Εδώ υπάρχει πλήρης συνένεση ότι δεν πρέπει να επιτρέπονται. Και αυτό αφορά τις εξαποστάσεως πωλήσει μέσω του διαδικτύου. Η έκθεση αντικτύπου λέει η Κομισιόν ότι δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχουν νόμιμες πωλήσει εξ αυτού του είδους, επομένως η Γενική Συνένεση είναι ότι μπορούν να απαγορευτούν. Κάποιοι συνάδελφοι θέλουν και περισσότερο. Θέλουν να απαγορεύσουν όλες τις πωλήσει μέσω διαδικτύου, ακόμα και μέσα στα κράτη-μέλη. Και εδώ η Κομισιόν μπορεί να σχολιάσει δεν ξέρω αν αυτό θα είναι νόμιμο ή όχι, αλλά μπορεί να μας πει η Κομισιόν. Τα καινοτόμα προϊόντα καπνού. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να εγκριθούν, τα κατημέλη θα μπορούν να ζητήσουν και να πάρουν μια έγκριση. Η Κομισιόν απλώς θα πρέπει να εφαρμόσει το γενικό σύστημα κοινοποίησης. Άλλοι λένε ότι πρέπει να αλλάξει ο τίτλος αυτής της, αυτού του τμήματος και να αναφέρονται ως λιγότερο βλαβερά καπνικά προϊόντα. Θα ήθελα και εδώ να υπάρχει κάποιο σχόλιο από αυτούς που έχουν καταθέσει αυτές τις τροπολογίες να μας εξηγήσουν γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί γίνονται αυτές τις τροπολογίες πολύ καλά. Ίσως οι συντάκτες τους μπορούν να εξηγήσουν καλύτερα. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα που περιέχουν νοικοτήνη. Είχαμε μια ειδική συζήτηση για τα θέματα αυτά. Οι τροπολογίες ποικίλουν όλο το φάσμα για τα προϊόντα με νοικοτήνη. Λένε ορισμένοι συνάδελφοι ότι αυτή, αυτό το νομοθέτημα δεν πρέπει να καλύπτει τα προϊόντα που περιέχουν νοικοτήνη. Άλλοι λένε ότι, ότι μόνο αυτά τα οποία έχουν μια, ένα ισχυρισμό για την ανθρώπινη υγεία θα πρέπει να υπόκεινται σε ρύθμιση. θέλουν να έχουν όρια ηλικία για τα τσιγάρα αυτά. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, εκτός αν υπάρχει μια διαδικασία έγκρισης για τα προϊόντα αυτά ειδική. Δεν ξέρω τι νομίζει η Κομισιόν για αυτά τα θέματα και τις τροπολογίες. Υπάρχουν επίσης πολλοί συνάδελφοι που θέλουν όλα τα προϊόντα που περιέχουν νοικοτήνη και τα πάτσες ε, και τα τσιγάρα να αναφέρονται ως φαρμακευτικά συσκευάσματα και δεν θέλουν η Κομισιόν να έχει δύο διαφορετικές κατηγορίες και οι τσίχλες επίσης. Επίσης τα ομοιοπαθητικά προϊόντα να υπάρχει ένα ελαφρό καθεστώς έγκρισης πιο λιγότερο επαχθές από το πλήρες καθεστώς. Δεν ξέρω και η Κομισιόν τι άποψη έχει για τα θέματα αυτά. Και υπάρχει μια τροπολογία από μένα και τον κύριο Φλόρεντς που είναι κάπως ενδιάμεση ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία έγκρισης για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά δεν πρέπει να θεωρηθούν φαρμακευτικά σκευάσματα, γιατί η οδηγία για τα σκευάσματα περιορίζει τη διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων. Υπάρχουν κάτι μέλη που επιτρέπουν αυτά τα προϊόντα να πουλούνται μόνο σε φαρμακεία, αλλά να πουλούνται οπουδήποτε αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για το θέμα των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Θα ήθελα να ξέρω την άποψη των συναδέλφων για όλα αυτά τα θέματα. Κάποιοι λένε πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σαν να είναι φαρμακευτικά σκευάσματα, άλλοι με καθόλου αυτό τον δρόμο. Από ό,τι ξέρω το Συμβούλιο, μάλλον θα θεωρήσει ότι όλα τα προϊόντα που περιέχουν νοικοτήνη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν φαρμακευτικά σκευάσματα. Αυτά λοιπόν πιστεύω ότι είναι τα κύρια θέματα. Υπάρχουν άλλες ίσονες τροπολογίες, κάποιοι συνάδελφοι να διευρύνουν αυτήν την ε, οδηγία για να απαγορεύσουν την πώληση σε συγκεκριμένους χώρους. Κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να είναι στα σούπερ μάρκετ, αλλά ούτε και στα μικρά καταστήματα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θέλουν να απαγορεύσουν τα, ε, προϊόντα που μιμούνται τα τσιγάρα, δηλαδή τα παιδικά παιχνίδια που είναι σαν τσιγάρα ή τα τσιγάρα τα οποία είναι απλώς γλυκά ή τσίχλες ή οτιδήποτε τέτοιο. Παλιά δίναν στα παιδιά για δώρο ένα πακέτο τσιγάρα που αντί για τσιγάρα είχε σοκολατάκια. Για κάποιους συναδέλφους αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά μπορούν να εξηγήσουν τις τροπολογίες τους αν θέλουν. Υπάρχουν άλλα θέματα λοιπόν για τα οποία δεν θέλω να αναφερθώ. Τώρα προτιμώ να ακούσω τις δικές σας απόψεις για τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ λέω Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή αυτή. Και τώρα να αρχίσουμε με τους κοιόδης συγητές Φλόρενς, Ντις, Καρούτα, Κένενεν, Όσοι, Ένδεσεν. Καλ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ την Λίντα Μακάβαν για τη συνεργασία του τελευταίους μήνες Όποιος διαβάσει τροπολογίες, περίπου 1300, θέλει μια εβδομάδα, δεν τις διάβασα όλες, αλλά όποιος τις ξεφυλίζει έστω, καταλαβαίνει ότι πάνε από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό να επιτευχθούν συμβιβασμοί. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είμαστε Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή. Ορισμένοι μπορεί να θεωρούν ότι είμαστε Επιτροπή Προώθησης της Οικονομικής Δραστηριότητας. Το καταλαβαίνω. Αλλά προς το παρόν ακόμη είμαστε Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών. Άρα πρώτη στην προτεραιότητα είναι η προστασία των καταναλωτών. Μπορεί να υπερβάλλει κανείς βέβαια. Ε, με εκπλήσει ε, η ευελιξία των ε, φιλελευθέρων. Ένας συνάδελφος φιλελεύθερος ζητάει να απαγορευτεί εντελώς η πώληση σιγαρέτων, ενώ ένας άλλος ε, επίσης φιλελεύθερος λέει ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα για αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει. Σας παρακαλώ, αναφερθήκατε σε έναν συνάδελφο Σας παρακαλώ, επιτρέψτε να συνεχίσετε να τηλεφωνάει. Όταν διάβασα τις τροπολογίες κάποιου συναδέλφου, ο οποίος έλεγε ότι είναι τραυματική η εμπειρία που είχε όταν διάβασε αυτήν την έκθεση, αλλά και εγώ είχα τραυματική εμπειρία όταν διάβασα, διάβασα τις τροπολογίες του. Εν πάση περιπτώσει, ας μην μπλέξουμε τις εφημερίδες τώρα. Θα πάρει ο συνάδελφος το λόγο μετά. Θα πάρει ο συνάδελφος το λόγο μετά. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η παρέμβαση ήταν αγένεια. Αγένεια. Θα ήθελα παρακαλώ πώς έχεις την ιδέα ότι ε, απλώς ε, ε είμαι εκπρόσωπος ενός λόμπι. Όταν κάνεις τέτοιες, ε, τέτοιους ισχυρισμούς θα ήθελα να μη είσαι πιο συγκεκριμένος. Θα δεν είναι δυνατόν να γίνουν τέτοια πράγματα. Πρέπει να παρεύει ο πρόεδρος. Τέσσερις ε, βουλευτές έχουν το ίδιο ακριβώς κείμενο υποβάλει. Εάν μου πείτε ότι και οι τέσσερις κατέληξαν αυτόνομα στο ίδιο ακριβώς κείμενο, τέσσερις, τέσσερις βουλευτές υπέβαλαν το ίδιο κείμενο. Αυτό λέξη δεν είναι δυνατόν να υποβάλλεται όλο το ίδιο κείμενο. Θα πρέπει να είστε λίγο πιο επιδέξιοι. Αλλά εντάξει, θα ακούσουμε αργότερα. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα που δεν καταλαβαίνω. Το τελευταίο της κυρίας Μακάβαν, ότι στο μέλλον όλα τα προϊόντα του καπνού θα πρέπει να απολούνται σαν παράνομα, δηλαδή να τα βγάζουμε από κάτω από, το, από τον κισέ. Ε, δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Τότε θα πρέπει και άλλα προϊόντα που μπορεί να είναι ε, επιβλαβή για την υγεία, όπως το γάλα και, το βούτυρο. Εν πάση και για το σνούς τώρα δεν θα πρέπει να είναι δικαιολογία ή μάλλον πρόσχημα για να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Αυτό δεν θα πρέπει να επιτρέψει και άλλες χώρες να ζητήσουν τέτοιες εξαιρέσεις. Δεν θα πρέπει να ε, ανοίξουμε αυτό το παραθυράκι. Δεν θα υποστήριζα λοιπόν εάν το σνους είναι σουηδική υπόθεση και πρέπει να μείνει τότε δεν χρειάζεται ευρωπαϊκός κανονισμός γι' αυτό. Θα το απέριπτα αυτό. Όμως είναι σαφές ότι ορισμένοι θέλουν απλή συσκευασία, το ξέραμε, και αυτό για μένα είναι υπερβολικό. Μπορούμε να συζητήσουμε βέβαια και για το μέγεθος των εικόνων και να διαφωνήσουμε ενδεχομένω γι' αυτό, θα μπορούσα να δεχθώ αυτά που λέει η Κομισιόν για τις συσκευασίε, εάν δεν είναι απλή συσκευασία. Δεν μου αρέσουν επίσης οι ιδιαίτερα μικρές συσκευασίε ε, ε, σιγαρέτων για πάρτι. Γιατί αυτά είναι πολύ ελκυστικά. Αυτό μας το δείχνουν ε, και τα στοιχεία για τις πωλήσει. και τα τσιγάρα slim, τα πολύ λεπτά τσιγάρα επίσης ε, είναι ιδιαίτερα ελκυστικά. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ πωλήσει τους ενώ πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν καθόλου τέτοιες πωλήσει. Ένα θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι κατά πόσο επιτρέπεται να μπαίνουν διάφορα πρόσθετα στα τσιγάρα. Εδώ και δεκαετίες η βιομηχανία μας κορυδεύουμε αυτό το θέμα. Πριν από 5-6 χρόνια ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Έπρεπε να μας ε, κάνουν εκθέσεις όχι ε, για ένα ή δύο συγκεκριμένα πρόσθετα, αλλά για 70 περίπου τέτοια ε, πρόσθετα που βάζουν. Θα, υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει κατά τη γνώμη μου θετικός κατάλογος και οι εμπειρογνώμονες να αποφασίσουν αν ε, το μεντόλ ή το, η ζάχαρη πρέπει να επιτρέπονται. Εγώ δεν ξέρω. Να μας πούν οι εμπειρογνώμονες. Θα ήθελα να μας πούν οι εμπειρογνώμονες. Όπως ξέρετε όταν καπνίζετε κοντά στη μύτη σας έχετε 800 βαθμούς ε, Κελσίου. Και στους 800 βαθμούς Κελσίου είναι ιδιαίτερα τοξική η ζάχαρη. Να μας τα πούν λοιπόν οι εμπειρογνώμονες. Εάν χρειάζεται τέτοια πρόσθετα στο τσιγάρο, τότε δεν θα αύξανα το ποσοστό μεντόλ, αλλά θα ήθελα να υπάρχει ένα νέο είδος καπνού. Αλλά εάν ο καπνός που καλλιεργούμε είναι τόσο κακής ποιότητας που δεν μπορούμε να το καπνίσουμε και το στέλνουμε σε άλλες χώρες και ε, οι άλλες αυτές χώρες ε, όπου έχουν περισσότερο ήλιο και τα καπνά εκεί λοιπόν είναι πιο όρημα και τα εισάγουμε ε, είναι ένας φαύλος κύκλος. Βεβαίως ένα νόστιμο πουρο θα έπρεπε να μυρίζει καπνό. Επίσης διαμεθοριακές πωλήσει είναι κακό πράγμα σίγουρα για τις εικόνες τώρα. θα μπορούσα να δεχτώ και εθνικές ρυθμίσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πλειοψηφία γι' αυτό εδώ. Αν πρέπει να είναι 75% τώρα του πακέτου οι εικόνες, θα μπορούσα να προτείνω ένα συμβασμό. Αυτοί που θέλουν 50% να είναι εικόνες, στην ουσία ε, θα δεχθούν και το 70%. Μπορούμε να το συζητήσουμε θα πρέπει να μελετήσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες ε, το επόμενο χρονικό διάστημα, να συγκρίνουμε και τι ακριβώς λέει ο κλάδος γι' αυτό και νομίζω ότι ορισμένοι εκνευρισμοί θα ηρεμήσουν. Πρόεδρος βεβαίως ε, έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις και για άλλες εκθέσεις. Βέβαια δεν μπορούμε να ελέγξουμε από πού προέρχονται οι τροπολογίες αλλά βεβαίως ορισμένες φορές μπορεί να δει κανείς ε, που υπήρξε η αρχική διατύπωση. Πρέπει να το συζητήσουμε. η Φρεντρίκ Ρίς ε, από πλευράς των φιλελευθέρων. Σας ευχαριστώ. Βλέπω πως η εκστατεία για τις ευρεκλαγές ε, του χρόνου έχει ήδη ξεκινήσει, τουλάχιστον στη Γερμανία. Εγώ για τα όσα μας απασχολούν σήμερα θα ήθελα εγώ να ε, ευχαριστήσω τώρα την εισηγήτρια και δεν είναι τυπικός, ε, τυπικά ευχαριστήρια, είναι τιτάνιο το έργο που έχει αναλάβει. Έχει συνεργαστεί και αν δούμε και πόσες νομοδοτήσεις περιμένουμε θα πρέπει να ξεκινήσει ήδη με τις συμβιβαστικέ και σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο εύκολο ούτε στο εσωτερικό των ομάδων. Βλέπουμε πόσο διαφορετικές και ποικίλε είναι οι ε, προτάσεις και οι θέσεις και δεν είναι και εύκολο ούτε με τις επιτροπές που είναι αρμόδιες για γνωμοδότηση γιατί από όσα μπόρεσα να διαβάσω ήδη και οι θέσεις που διαγράφονται εκεί στην ΙΜΚΟ αλλά και στην ε, Επιτροπή Βιομηχανίας αλλά και στην ε, η ε, ε, ε, νομική επιτροπή οι απόψεις είναι αποκλίνωσες και σίγουρα θα χρειαστεί χαλάρωση όπως το θέμα της συσκευασία, το μέγεθος των προειδοποιήσεων για την υγεία, τα λεπτά τσιγάρα και το καθεξής, πολλά ζητήματα και εν γέννη πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τις βασικές προόδους που περιλαμβάνονται σε αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Ήδη θα ήταν μεγάλη νίκη. Προφανώς για να δούμε λίγο τα περισσότερα σημεία και τις προτεραιότητές μας, να σας πω ότι σίγουρα θέλουμε να διατηρηθεί και η απαγόρευση για των αρωμάτων και των προσθετικών, παράγραφος, ε, άρθρο 6, παράγραφη 3 και 4, βανίλια, ε, καραμέλα, τα λοιπά Τουλάχιστον αυτό για την ομάδα των φιλελευθερών, να σας το λέω ότι ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να εκφραστούμε ομόφωνα. Και εδώ λοιπόν εμείς συμπεριλαμβανομένουμε και τη μεντοθόλη, γιατί η Λίντα Μακάβαν εξήγησε γιατί είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η απαγόρευση. Επίσης σημαντικό σημείο είναι το να επιτεθούμε στις πιο καρκινογόνες για την υγεία είναι το αντικείμενο μιας τροπολογίας που κατέθεσα εγώ για το άρθρο 5 μαζί με την Κόριν Λεπάζ που στόχο έχει να προτείνει ένα κατάλογο για τα πρότυπα που υπάρχουν στη ΣΥΠΑ για τις ουσίες της πιο επικίνδυνες ανακατηγορία καπνού. Δημιούργησα λοιπόν δύο παραρτήματα που στόχο έχουν να απαριθμίσουν καταρχήν αυτές τις ουσίες πριν να προβλεφθεί και ο περιορισμός τους σε, σε μια δεύτερη φάση και θα ήθελα να διευκρινίσω πως αυτός ο κατάλογος, αυτό η απαρίθμηση δεν είναι ασύμβατο με, τη θετική, με το θετικό κατάλογο κατάλογο που αναφέρθηκε επίσης και για τον οποίο από ό,τι κατάλαβα έχει μια κάποια συμπάθεια η συγγήτρια έχει κατατεθεί από διάφορους συναδέλφους και καθώς επίσης και οι 422 και 424 τροπολογίες που μέσα στο πλαίσιο της μέγα νομοθεσίας REACH που κατατέθησαν από τον κύριο Φλόρενς και που όντως ε, οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι προφανές ότι δεν θα υποστηρίξουμε φυσικά την πολύ πιο σκληρή γραμμή, την πολύ ρηξικέλευτη γραμμή που είναι αυτή που υποστηρίζει μια ολόκληρη ομάδα συναδέλφων, Βίλμοντ, Σλίτερ, ε, κάποιοι ε, ε, Βουλευτέ τη ομάδα μου πιστεύω πω θα πρέπει να είμαστε συνεπεί. Είναι αυταπάτη να θέλουμε να καταστήσουμε τον καπνό ένα τελείω ακίνδυνο προϊόν καθόλου βλαβερό και καθόλου τοξικό. Συνέπεια θέλουμε, όπω είπαμε, ναι, μηδενική ζημιά, μηδενική βλάβη θα ήταν αυτή η προσέγγιση των πιο ε, ριζοσπαστικών φιλελευθέρων όπως ο Τουάν Μάντερς στην τροπολογία 444. Εκείνος εντάξει το είπε. Κανονικά θα πρέπει να απαγορευτεί ε, το κάπνισμα. Ε, να πει κανείς ότι ο καπνός είναι καραμέλα ή γλυφιτζούρι, δεν είναι γλυφιτζούρι. Οι φιλελεύθεροι που εγώ αντιπροσωπεύω λοιπόν δεν θα υποστηρίξουν ούτε, και το λέω και στην εισηγήτρια, εκτός και αν υπάρξει κάποια εξέλιξη στις συμβιβαστικέ, είναι οι 1250 που υπέβαλαν η εισηγήτρια αλλά και το ΕΛΚ, δηλαδή τα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά τσιγάρα, που μεγάλη συζήτηση και εκεί, αυτά που περιέχουν νοικοτήνη, γιατί είπαμε ότι από συζήτηση σε συζήτηση και από ραντεβού στο, σε ραντεβού και από ακρόαση σε ακρόαση, είναι σημαντικό να στηρίξουμε μια θέση που θα καθιστά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα λιγότερο προσβάσιμα από ό,τι τα τσιγάρα. Ε, για να μου εξηγήσετε θέλετε χιλιάδες χρόνια για να με πείσετε πώς θα συνεχίσουμε να πουλάμε πουθεν, παντού τον ε, καπνό, τα τσιγάρα, ενώ το ηλεκτρονικό τσιγάρο το οποίο μειώνει του κινδύνου θα είναι προσιτό με πολύ πιο περίπλοκο τρόπο και μόνο στο φαρμακείο. Για, κατά την άποψή μου κάτι τέτοιο δεν είναι ε, λογικό. Υπάρχουν εκατομμύρια χρήστες αυτών των ατμοποιητών ε, στην Ευρώπη. Ε, πιστεύω πως δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Είναι ακατανόητο κάτι τέτοιο αυτή η πορεία προς την αποκλειστικότητα στα φαρμακεία. Είναι, ενώ το τσιγάρο είναι διαθέσιμο παντού και το ηλεκτρονικό τσιγάρο να απαγορεύεται και να υπάρχει μόνο, να διατίθεται μόνο στα φαρμακεία. Αδύνατον για μας. Όσον αφορά τώρα την ευθυγράμμιση με την πρόταση της Κομισιόν και της επισηγήτριας σύμφωνη για την απαγόρευση των εξαποστάσεων πωλήσεων κυρίως στο ίντερνετ, ε, αδειοδότηση κυρίως ε, για τα νέα προϊόντα καπνού, για τις διαφημίσεις για τους νέους, ας πούμε, διωρεάν διανομή τσιγάρων κτλ. Απαγόρευση των αρωματικών ουσιών, το είπα, και για τη μενθόλη. Για το σνούς ε, συμφωνούμε για ένα είδος status quo, σύμφωνοι με την εξαίρεση για τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Και μάλιστα θα τίναμε και να τους αφήσουμε να διατηρήσουν και τα αρώματα που χρησιμοποιούν. Εγώ δεν έχω ποτέ καπνίσει τους ή άλλους, ούτε έχω χρησιμοποιήσει το σνούς και δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά φαντάζομαι ότι χωρίς άρωμα θα είναι πραγματικά αδύνατο να το χρησιμοποιήσει κανείς. Τώρα για τη σίσα, για τους ναργιλέδες. Ε, και εδώ να πω και είναι γνωστό ότι είναι μόδα στους νέους, τους ελκύει και όπως είπαμε οι νέοι είναι το βασικό μας στόχος για την προστασία. Είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε λοιπόν και με τον αργυλέ. Το θέμα της συσκευασία ε, συμφωνούμε γέννη να ακολουθήσουμε την πρόταση της Κομισιόν, 75% γύρω από αυτό δεν ε, είμαστε απόλυτοι για τις τροπολογίες που είναι στο 65, 70 ή ακόμα και 80%. Θα έλεγα απλά ότι συμβολικά το να είμαστε κάτω από τη φιλοδοξία της Κομισιόν δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Εγώ που είμαι από το Βέλγιο είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη και είμαστε πάνω από το 70% και είναι πιο εύκολο για μένα ε, Βέβαια, οι συνδυασμένες απόψεις των, είναι ούτως ή μόνο για δέκα κράτη ε, δεκτές. Και να αναφέρω και τα όσα είπε ο κύριος ε, Τουάν Μάντερς ε, με, με ενδιαφέρουσα ιδέα, γιατί ίσως στην πρωτοτυπία θα βρούμε και τη λύση. Πραγματική λύση δεν είναι το δικό μας χέρι είναι η τιμή και επειδή ακριβώς δεν είναι δικό μας θέμα Ο Μάντερς λοιπόν προτείνει να διπλασιαστεί το βάρος του πακέτου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ένας νεαρός καπνιστής έχει δύο εμπόδια. Είναι βαρύ και είναι και πολύ ακριβό για ένα νέο. Είναι πραγματικό το εμπόδιο λοιπόν και δεν είμαι αθώα λέγοντάς το αυτό. Θέλουμε να συμβουλέψουμε τους υπουργούς μας, υπουργούς υγείας, υπουργούς κοινωνικών, κοινωνικής πρόνοιας, υπουργούς οικονομικών. Εξακολουθώ να βρίσκω παράδεκτο που ε, τα τσιγάρα κοστίζουν, ο καπνός μάλλον κοστίζει μια φορά, δύο φορές λιγότερο από τη, το καπνό στη Βρετανία ή αλλού ε, και ότι στην ουσία εμείς εξάγουμε προϊόντα καπνού. Αυτή είναι η ουσιαστική συζήτηση. Ευχαριστώ. Η Σάτου Χάση έχει <clears throat> το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να ευχαριστήσω και το, την εισηγήτρια με την οποία μπορώ να συμφωνήσω σε πάρα πολλά θέματα. Ήταν μια μεγάλη ευχαρίστηση να ακούσω τον ε, Καλ Χάιντς Φλόρεντς από το ΕΛΚ να επικρίνει τους συναδέλφους οι οποίοι απλώς μεταφέρουν αυτολεξή τις τροπολογίες που έρχονται από, την, από τις βιομηχανίες τσιγάρων. Έχω τρία, τέσσερα θέματα για τα οποία θα ήθελα να σταθώ. Καταρχήν η απλή συσκευασία. Εγώ νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη η κίνηση προς την απλή συσκευασία. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το κάπνισμα είναι από τους μεγαλύτερους φωνιάδες. 700.000 άτομα σκοτώνει κάθε χρόνο στην Ευρώπη, του σκοτώνει πρόωρα. Και θα πρέπει, δεν θα μπορεί να είναι, δεν πρέπει να είναι δυνατόν να μπορούμε να εμπορευόμαστε ένα τέτοιο φωνικό προϊόν σε πολύχρωμα και ευχάριστα πακέτα. Η συσκευασία είναι το πιο ουσιαστικό εργαλείο επικοινωνίας των ε, σιγαροβιομηχανιών προς τον καταναλωτή. Γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε την απλή συσκευασία. Ένα δεύτερο σημείο. Οι προσθετικές ουσίες. Η Λίντα εξήγησε ήδη πολύ καλά γιατί οι προσθετικές ε, ουσίες με τις οποίες περιλαμβάνουν και τις αρωματικές ουσίες και τη μενθόλη θα πρέπει να απαγορευτούν όλες. Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι η σύμβαση πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζητά από όλες τις συμβαλόμενες πλευρές να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τις προσθετικές ουσίες που κάνουν πιο εύγευστα τα καπνικά προϊόντα. Το να απαγορεύσουμε λοιπόν τις αρωματικές ουσίες ακριβώς σημαίνει ότι ακολουθούμε αυτά τα οποία έχουμε δεχτεί μέσα στη σύμβαση πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η δική μας πολιτική ομάδα έχει προτείνει να καταρτιστεί ένας θετικός κατάλογος που αναφέρθηκε σε αυτόν η Λίντα Μακάβεν. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι μόνο συγκεκριμένες ουσίες, οι οποίες δεν είναι αρωματικές προσθετικές ουσίες ή κάνουν με άλλο τρόπο πιο εύγευστα ή πιο αλκυστικά τα τσιγάρα, μόνο αυτές οι ουσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην σύνθεση των τσιγάρων και επίσης ουσίες οι οποίες δεν είναι αφέ αυτού βλαβερές. Θα υπάρχουν λοιπόν αυτά τα κριτήρια και μια διαδικασία λήψης απόφασης για τις ουσίες αυτές και όλα αυτά βρίσκονται στην τροπολογία μας 583. Μια τρίτη παρατήρηση, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Νομίζω ότι χρειάζονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως ένας τρόπος για τους καπνιστές να σταματήσουν βαθμία το κάπνισμα. Αλλά οι μελέτες που μας έχουν παρουσιαστεί δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Δεν είναι ούτε ασφαλή ούτε αξιόπιστα. Θα είχε λοιπόν νόημα να τα ταξινομήσουμε, να τα κατατάξουμε στα φαρμακευτικά προϊόντα όπως προτείνει η Κομισιόν. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πρέπει να πολλούνται μόνο στα φαρμακεία. Αυτό εναπόκειται στα κράτη-μέλη να το ρυθμίσουν. Δεν είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να αποφασίζει κάθε κράτος μέλος πού μπορούν να απολούνται αυτά τα προϊόντα, αν μπορούν να απολούνται πέραν των φαρμακείων και σε άλλα καταστήματα. η απέτηση έγκρισης ως φαρμακευτικών προϊόντων δεν σημαίνει ότι εμείς θα περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα των ε, ηλεκτρονικών τσιγάρων και θα πολλούνται μόνο στα φαρμακεία. Αλλά πρέπει να είμαστε ισοδίκαιοι και έναντι των βιομηχανιών και να επιτρέψουμε ένα ε, μεταβατικό διάστημα. Και εδώ έχουμε προτείνει τέσσερα χρόνια για αυτή τη μεταβατική περίοδο. Ένα τέταρτο σημείο στο οποίο δεν έχει σταθεί κανείς ακόμα αλλά για το οποίο εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογίες και θα ήθελα να το συζητήσουμε στο πλαίσιο αυτό, είναι το θέμα της περιεκτικότητας πολωνίου μέσα στα τσιγάρα. Αυτό φυσικά δεν γίνεται θεληματικά. Αλλά το πολονίο περιέχεται ήδη στον καπνό ως προϊόν αποσύνθεσης του ουρανίου. Ραδιενεργής αποσύνθεσης του ουρανίου. Αυτό είναι κάτι που προέρχεται από τα λιπάσματα που περιέχουν ουράνιο. Όταν καίγεται το τσιγάρο, το πολόνιο μπαίνει στα, στους πνεύμονές μας, είναι ε, εκπέμπει ακτίνες α που είναι το πιο επικίνδυνο ε, πιο επικίνδυνη μορφή ραδιενέργειας. Το να καπνίζει κανείς 20 τσιγάρα την ημέρα είναι το αντίστοιχο του να έχει κάθε χρόνο 200 ε, ακτινογραφίες τώρα κατό χρόνο. Είναι σημαντική λοιπόν η έκθεση σε ραδιενέργεια και υπάρχουν απλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε το, το, την περιεκτικότητα σε πολώνιο του καπνού. Προτείνω να υπάρξει λοιπόν ένα όριο για την περιεκτικότητα σε πολώνιο των ε, τσιγάρων. Ευχαριστώ. Η Αν Ρόσπαχ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνω το λόγο εξ του Μάρτιν Κέλεναν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω καταρχήν την εισηγήτρια για την έκθεσή της και για την πολύ καλή συνεργασία που έχει κρατήσει με τους κύριους εισηγητές. Προσπαθώ να είμαι σύντομη. Ο κύριος Κάλανεν έχει ορισμένα μονάχα σημεία που θέλει να θίξει. Το πρώτο είναι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Εδώ μας ανησυχεί η προσέγγιση της εισηγήτριας στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και ο αριθμός των τροπολογιών που έχουν αναφερθεί. Αναφέρθηκε σε πάρα πολλέ τροπολογίες, δεν θα διαβάσω τους αριθμούς τους, αλλά τα έχω εδώ όλα αυτά, στοιχεία αν θέλετε. Σε ένα ιδανικό κόσμο κανείς δεν θα ήταν εξαρτημένος από τον καπνό. Στον πραγματικό κόσμο όμως υπάρχουν εκατομμύρια Ευρωπαίων που είναι εθισμένοι και εξαρτημένοι από τα καπνικά προϊόντα. Και όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, οι μισοί από αυτούς θα πεθάνουν ακριβώς λόγω αυτής της εξάρτησης από τα καπνικά προϊόντα. Νομίζουμε ότι η συγγήτρια δεν καταλαβαίνει ακόμα πόσο ομές είναι οι τακτικές αυτές μείωσης της πρόσβασης σε ηλεκτρονικά σιγάρα. Ο δικός μας σκιώδης εισηγητής είπε ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψει κανείς τον πρόωρο θάνατο από κάπνισμα. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι μέχρι το 2017 το αργότερο η Κομισιόν θα πρέπει να προβεί σε μια πλήρη ανάλυση κόστους ωφέλους και ανάλυσης κινδύνων υγειονομικών για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Γιατί μιλάμε για εκατομμύρια ζωές οι οποίες διακυβεύονται. Είναι απαραίτητο να έχουμε την καλύτερη δυνατή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Για την τυποποίηση τώρα της ε, συσκευασίας και της προειδοποίησης για θέματα υγείας. Αναγνωρίζουμε ότι εδώ ο στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση της δημόσιας υγείας. Αλλά μας ανησυχεί ακόμα ο αντίκτυπος αυτής της νομοθεσίας στην εμπορία, στον ανταγωνισμό των διαφόρων ειδών τσιγάρων. Υπάρχει η εμπειρία της Αυστραλίας και υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν μια τέτοια ρύθμιση απλής συσκευασία, αλλά αυτό νομίζω ότι αντιβαίνει των κανόνων της αγοράς. Επομένως, μια νομοθεσία που αφορά την ενιαία αγορά ε, δεν θα πρέπει να αφαιρέσει οποιαδήποτε δυνατότητα να προωθούνται συγκεκριμένες μάρκες τσιγάρων. Υπάρχουν περιορισμοί βέβαια. Πολλοί για την αγορά χαμικών προϊόντων δεν νομίζουμε ότι περαιτέρω περιορισμοί θα βοηθήσουν τη δημόσια υγεία. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι με τον τρόπο αυτό δεν θα υπονομεύσουμε τη δυνατότητα συμφωνίας, επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση. Και προσωπικά θα ήθελα να προσθέσω το εξής ότι έχουμε τις εικόνες αυτές τα πακέτα τσιγάρων, αλλά οι περισσότεροι καπνιστές βάζουν σε μια θήκη το πακέτο τσιγάρων τους και δεν βλέπουν αυτές τις εικόνες. Και για το σνούς, και αυτό είναι το θέμα της εξαίρεσης για τη Σκανδιναβή, δεν είναι μόνο σκανδιναβικό θέμα το σνούς. Και οι Φινλανδοί και οι Δανείοι και οι Νορβηγοί που οι Νορβηγοί τελευταίοι δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοί χρησιμοποιούν το πολύ σνούς, βέβαια δεν έχει την ίδια έκταση χρήση του όπως στη Σουηδία. Πιστεύουμε λοιπόν, ή πιστεύει μάλλον και ο συζητητή μας, ότι θα πρέπει να αφήσουμε και κάποιο περιθώριο για τις χώρες αυτές να χρησιμοποιούν το σνους, γιατί υπάρχει μια μακραίωνη παράδοση και πρέπει να παραμείνει νόμιμο το σνους στις χώρες αυτές. Και τέλος, ανεκδοτολογικά, ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορούμε να έχουμε και καφεΐνη στον καφέ που πίνουμε στην Επιτροπή μας και ελπίζω ότι δεν θέλει κανείς να απαγορεύσει την χρήση καφέινης στον καφέ μας. Αγαπητή Άννα, λέει ο πρόεδρος, Ορισμένοι συνάδελφοι έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο και έχουν βάλει το Union Jack την αγγλική σημαία πάνω στα, στα φλιτζάνια τους. Ο κύριος Ρώση έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ συνεχίζω να είμαι πολύ επιφυλακτικός και επικριτικός για αυτό το κείμενο. Ε, της Κομισιόν αλλά και για αυτή την στάση Ταλιμπάν της εισηγήτριας. Δεν μπορεί αύριο να έρθει αύριο κανείς να μας πει ε, ότι η καφεΐνη βλάπτει αύριο μεθαύριο και ξαφνικά να πρέπει να τιμωρήσουμε και αυτούς που πίνουν πολλούς καφέδες. Αυτό το κείμενο λοιπόν, ο φόβος μου είναι ότι στην ουσία θέλει να ε, τακίσει τον καπνιστή. Εκεί δηλαδή όπου ο πολίτης, εντάξει, είμαι υπέρ της απαγόρευσης της πώλησης προς τους ε, ανήλικους, δηλαδή ένας ενήλικο πολίτης θεωρείται ότι δεν μπορεί να αποφασίσει. Θέλει λέει, να αυτοκτονήσει από μόνος του για να... και δεν μπορεί να αποφασίσει τι να κάνει. Και εμείς ο νομοθέτης πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτό το βίτσιο του να γίνει ε, έγκλημα, ε, ποινικό αδίκημα. Δεν μπορεί να βρει ούτε ένα αγαπημένο του μάρκα, ούτε συγκεκριμένο καπνό, γιατί εμείς αποφασίσαμε ότι δεν πρέπει να καπνίσει γιατί του κάνει κακό. Μα αυτό δεν είναι σωστό, γιατί αύριο μεθαύριο η καφεΐνη είπαμε μπορεί να μας πει να καταργήσουμε ας πούμε, τα επικίνδυνα αθλήματα γιατί βλάπτουν ή τα λιπαρά γιατί βλάπτει, το αλκοόλ γιατί βλάπτει. Ε, εντάξει, τότε θα τα καταργήσουμε όλα. Είδα εκείνο το, την κάρτα που σπονσοράρει η συγγήτρια για ένα συνέδριο Μα εκεί πια δεν, δεν, υπάρχει πια ελευθερία επιλογής. Εμένα με φοβίζει κάτι τέτοιο. Ε, αγαπητοί φίλοι. Εντάξει, να δώσουμε την κατάλληλη ενημέρωση, ναι, Σύμφωνη. Στην Ιταλία πάντω σίγουρα δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται στι άλλε χώρε τη ε, Ένωση. Σίγουρα πάντω στην Ιταλία δεν υπάρχουν ε, στο σχολείο ε, μαθήματα που να εξηγούν τι βλαβερέ συνέπειε του καπνού κτλ. Ελάχιστα πράγματα γίνονται. Να ενημερώσουμε, ναι, και από τη στιγμή που είναι κανεί ενήλικο να μπορεί να διαλέξει ο ίδιο να επιλέξει τι θέλει να κάνει χωρί να δημιουργεί πρόβλημα και για του άλλου δίκαιο να αποφεύγεται, να απαγορεύεται μάλλον το κάπνισμα σε κλειστού χώρου και να απαγορεύεται να ενοχλεί του άλλου καπνίζοντα. Αλλά ένα άνθρωπο ενήλικα και ενήμερο που επιλέγει παρόλα αυτά να καπνίζει, δικαίωμά του δεν του το απαγορεύει πλέον ο νομοθέτη. Ή άμα θέλει να καπνίζει μικρό, λεπτό, χοντρό, ε, άσπρο, μαύρο τσιγάρο, δική του δουλειά. Εμεί τι σχέση έχουμε, γιατί μπορούμε να λέμε στου ανθρώπου ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Και υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι λέει πρέπει να απελευθερώσουν με τα ελαφρά ναρκωτικά. Δηλαδή Γιατί αυτά είναι καλά για την υγεία μήπως. Εκείνα εκεί να απελευθερωθούν. Ε, νομίζω πως έτσι ανοίγουμε ένα μέτωπο περιορισμού της ελευθερίας, της προσωπικής ελευθερίας. Για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και εγώ ανησυχώ για αυτή την υπόθεση, γιατί δεν είμαι και τόσο βέβαιος ότι είναι και τελείως αυλαβής. Και επειδή εγώ ε, είμαι αντίθετο στο να θεωρηθούν ε, ε, φαρμακευτικά προϊόντα. Στι περισσότερε πτώσεις οι άνθρωποι που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, όταν θέλουν να σταματήσουν τσιγάρο, το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι υποκατάστατο του τσιγάρου δεν σταματάνε να καπνίζουν, χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο ει αντικατάσταση, μάλλον υποκατάσταση του κανονικού τσιγάρου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποιο ε, ε, προσθετικό μέσο, κάποιο πρόθεμα, ε, γιατί δεν έχει νόημα. Είναι ένα υποκατάστατο του τσιγάρου, είναι κάτι διαφορετικό, αλλά σίγουρα δεν είναι κάποιο ιατρικό προϊόν. Τώρα, εκείνο το κομμάτι που μιλάει για τι εσωτερικέ πολιτικέ του Κοινοβουλίου που τονίζει πολλέ από τι αμφιβολίε που εγώ αναφέρω, α πούμε αντίκτυπο στην εθνική οικονομία και στην απασχόληση. Για παράδειγμα, εμεί διευκρινίζουμε ποια είναι η πραγματική επιρροή στου κανόνε Διεθνού, εμπορίου, τον κίνδυνο τη αύξηση του λαθρεμπορίου λέει επίση αλλά αναφέρει και ότι δεν είναι σαφή ε, ο πραγματικό αντίκτυπο ε, τη τροποποίηση αυτού του πακέτου. Η ίδια μελέτη που έκανε οι του Κοινοβουλίου αναφέρουν ε, αμφιβολίε για τα όσα προτείνει η Κομισιόν σε σύγκριση με τα όσα προτείνουμε εμεί. Εγώ επαναλαμβάνω ότι η προσωπική ελευθερία πρέπει να είναι κυρίαρχο δικαίωμα για όλου του πολιτικού. Δεν μπορούμε εμεί να ε, υπαγορεύουμε σε ενήλικε και ενήμερου ανθρώπου τι να κάνουν. Η συνάδελφο Άντερσεν, που είναι σκιώδη ε, τη ε, ΓΚΟΕ. Α, θα γυρίσει από τη Ρέγκη, καλώς. Θα έρθει σε λίγο. Να διαβάσω το κατάλογο των ομιλητών που έχουν εγγραφεί. Αν κάποιος ε, δεν είναι, Ζέμπα, Ζάμα, Κράμα, Λίζα, Ατρόση, Ούλματ, Περίλο, Ρέγγις, Μελάνια, Κρίστοφα Φιέλνα. Ε, ξέχασα κάποιον? Όχι. Ωραία. η συνάδελφος ε, Γκαρντίνη, βεβαίω. Θα πρότεινα να δώσουμε τρία λεφτά στον καθένα για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Για να έχει ο καθένας ε, τη δυνατότητα να εκφραστεί για αυτό το σημαντικό θέμα. Ζήμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα και ιδιαίτερα την εισηγήτρια, του Σκιώδης, ε, τη γραμματεία που αντιμετώπισε 1.300 ε, τροπολίες. Ξέρω ότι δύσκολο είναι. Ως κοινοβούλιο έχουμε να παίξουμε ε, το ρόλο μας ως νομοθέτες και είναι δικό μας θέμα να καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτό το προϊόν στον κόσμο, είναι πραγματικότητα, πρέπει να το κάνουμε όσο πιο ασφαλές γίνεται γιατί ε, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως ε, πολιτικοί για θέματα υγείας. Βεβαίως ε, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κράτος δεσμοφύλακα, θέλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να μειωθεί η χρήση τσιγάρων, αλλά και για να είναι ασφαλέστερο αυτό το προϊόν. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η σύμβαση που υποχρεώνει όλα τα κράτη και υποχρεώνει και τον κλάδο ιδιαίτερα για τα προσθετικά. Πρώτον, να είναι πιο διαφανής και δεύτερον, να επιτρέπονται μόνο αν είναι ασφαλή. Γι' αυτό υπέβαλα τις τροπολογίες 94-69 ε, με το θετικό κατάλογο. Είναι σημαντικό νομίζω αυτό για να ε, υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Για τον κίνδυνο της, ε, του καπνίσματος βεβαίως είναι πολύ επικίνδυνα για τα παιδιά και τις εγγύους, γι' αυτό υπέβαλα τροπολογίες όπου αναφέρομαι σε αυτούς τους κινδύνους. Γιατί υπάρχει μια διαφορά αν ε, αποφασίζει κάποιος να καπνίσει ε, από τη μία και αν επιβάλλει τον καπνό ε, θίγοντας άλλους. Βεβαίως υπάρχουν αρκετές μελέτες που καταδεικνύουν ότι οι εικόνες παίζουν ε, ρόλο για να περιορίσουν το τσιγάρο. Και έχω κάποιες αφιβολίες εάν είναι σωστή η αντιμετώπιση της Κομισιόν ε, για το θέμα αυτό. Πρέπει να δούμε πώς ε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο το μέσο αυτό για να προωθήσουμε την υγεία. Κάτι άλλο Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλο συμφέρον, ε, πολλά πάθη, αλλά νομίζω είναι οριακός ο τρόπος με τον οποίο ο κλάδος επιχειρεί να μας ασκήσει πιέσεις. Το διαπίστωσα. Θα πρέπει να καλέσουμε τον κλάδο να ε, παίζει με ανοιχτά χαρτιά και οι εθνικές αρχές να παίξουν το ρόλο τους σε αυτή την κατεύθυνση γιατί αλλιώ ε, θα έχει αρνητικές επιπτώσει και για τον κλάδο αυτό η εξέλιξη της εξέτασης του θέματος. Κράμερ. Συγγνώμη, η κυρία Ζώμα. Ρενάτε Ζώμα. Δεν έχω αλλάξει όνομα, λέει η κυρία Ζώμα. Κοιτάξτε, ε, αναφερόμαστε μόνο σε νόμιμα προϊόντα μέχρι στιγμή. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γι' αυτό κάποιες προτάσεις τις ε, βλέπω κάπως υπερβολικές βεβαίως τα προϊόντα να γίνουν ασφαλέστερα. Και εγώ δεν θέλω να αρχίσουν να καπνίζουν οι νέοι. Αλλά τι ρόλο παίζουν οι νόμοι για την προστασία των νέων που έχουμε στα κράτη-μέλη. Πρέπει να τηρούνται καλύτερα. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό αφορά, αφορά και άλλα, για παράδειγμα, ε, προϊόντα, όπως ε, το ενόπνευμα. Δεν μπορούμε όλα να τα ρυθμίσουμε με ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Είμαστε σε συνθήκες κρίσης. Είναι κάπως κοινικός λοιπόν να γράφεται, όπως λέει η Κομισιόν, ότι θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας από τις προτάσεις μας. Αλλά θα δημιουργηθούν κάποιες νέες. Πού θα δημιουργηθούν κάποιες νέες θέσεις. Θα ήθελα να μάθω. Πού θα δημιουργηθούν με αυτή την ε, πρόταση νέες θέσεις εργασίας. Και όσοι θα χάσουν τις θέσεις εργασίας τους είναι καταναλωτές. Είμαστε προστασία, είμαστε επιτροπή καταναλωτών. Δεν θα πρέπει, επειδή είμαστε επιτροπή καταναλωτών, να θεωρούμε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για κανένα άλλο θέμα. Έχουμε ευθύνη για όλους μας τους πολίτες, τους οποίους εκπροσωπούμε. Για τις θέσεις εργασίας τους. Μιλάμε για νόμιμα προϊόντα. Η, Είναι λάθος αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα χνηλασιμότητας. Είναι υπερβολικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Ε, που κατόπιν ε, ε, αποθηκεύουν και πολλούν τσιγάρα είναι λάθος και η απλή συσκευασία νομίζω είναι λάθος δεν θα προστατεύσει από απομιμήσεις αντίθετα θα τις ευνοήσει θα πρέπει να επιτρέψουμε οι εταιρείε να βάζουν και στα τσιγάρα και στα πακέτα τα σήματα αυθεντικότητας γιατί εάν υπάρξει ε, απομίμηση θα ε, τίθεται εν κινδύνο ε, η υγεία των καταναλωτών. Μπορούμε να συζητήσουμε για διαδικασία έγκριση των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Τι θα γίνει με τις πίπες όμως και με το ΣΥΣΑ. Δεν είναι ακίνδυνα. Και αυτά είναι προϊόντα από τα οποία αρχίζουν να καπνίζουν οι νέοι. Για τις αρωματικές ουσίες είναι λάθος η γενική απαγόρευση. Πρέπει να προσέξουμε. Εάν εξαιρέσουμε το σνους, αυτός ε, ε, ε, το σνούς και όλη αυτή όλα αυτά τα είδη καπνού τα οποία τα βάζουμε στη μύτη μας ζουν μόνο αν έχουν και αρωματικές ουσίες και δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Όπως είπε η Μακάβεν, το θέμα που μας απασχολεί είναι η κατεξοδότηση πράξης. Είναι τόσο πολλές και οι τομείς που καλύπτουν είναι υπερβολικοί. Αυτό ε, οδηγεί σε αποδυνάμωση των αρμοδιοτήτων των Ευρωπαίων συνομοθετών. Ε, δίνει πλήρη εξουσιοδότηση στην Κομισιόν να ε, εισαγάγει μόνη της όλες περαιτέρω τροποποιήσεις του κανονισμού στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε για καθαρά τεχνικά θέματα της κατεξοδότηση πράξεις, αλλά αυτή η μαζική εισαγωγή τους είναι ξεδιάντροπη από πλευράς Κομισιόν και δεν θα πρέπει να την επιτρέψουμε. Ωραία. Ωραία. Ακολουθεί το λόγο η κυρία Άντερσεν από την ΚΟΕ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την επίοικη σας και ευχαριστώ και πάλι την Λίντα Μακάβεν για την πολύ σκληρή εργασία της λυπάμαι που χρειάστηκε να φύγω ε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έπρεπε να πάω στην Επιτροπή Ρέτζι. Έχουμε 1.360 τροπολογίες, ξέρω ότι πολλοί από τους ε, συναδέλφους βλέπουν τη δυσκολία του θέματος αυτού. Είναι σαφές ότι οι καπνοβιομηχανίες έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο για την άσκηση πιέσεων και λόμπινγκ αλλά χάρηκα που είδα κάποιε τροπολογίε από συναδέλφου που μοιάζουν με τι δικέ μου, που έχουν σαν στόχο να προστατεύσουν την ε, υγεία και τη ζωή των συμπολιτών μας και όχι τα θησαυροφυλάκια των εταιριών. Το θέμα της ε, τυποποιημένη συσκευασία έχει συζητηθεί ήδη, αλλά θέλω να τονίσω και μερικέ σημαντικέ εξελίξει που έχουν ε, λάβει χώρα στην Ιρλανδία, στη χώρα μου αυτή τη βδομάδα. Αναφέρθηκε ότι ο Έντα Κένι, ο Πρωθυπουργό και δύο από τους ε, υπουργού του έχουν κάνει μια συμφωνία με τις καπνοβιομηχανίες. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Και αναφέρθηκε ότι με τον τρόπο αυτό υπήρξε η κίνηση προς 100% τυποποιημένη συσκευασία. Έτσι η Ιρλανδία θα γίνει η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δεύτερη στον κόσμο μετά την Αυστραλία που θα εφαρμόσει αυτή την τυποποιημένη απλή συσκευασία. Αυτό θα δώσει και ένα σημαντικό προηγούμενο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα για τις συζητήσεις που γίνονται και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των αραματικών ουσιών, η Κομισιόν επιτρέπει, θέλει να επιτρέψει ορισμένες αρωματικές ουσίες εφόσον δεν δημιουργούν τις λεγόμενες χαρακτηριστικές αρωματικές γεύσεις. Εγώ υποστηρίζω μια πλήρη απαχώρευση των προσθετικών ουσιών που δεν έχουν καμιά θέση στην παραγωγή τσιγάρων και αυτό περιλαμβάνει οποιαδήποτε προσθετική ουσία μπορεί να κάνει πιο ελκυστικά τα τσιγάρα. Πιστεύω ότι οι προτάσεις της Επιτροπής είναι δύσκολες να εφαρμοστούν στην πράξη και αυτό το οποίο έχει ονομάσει Κομισιόν ανεξάρτητες ε, ε, ομάδες ελέγχου δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν καλά. Ο στόχος λοιπόν πρέπει να είναι να μην έχει μια ανεξάρτητη γεύση το καπνικό προϊόν εκτός από αυτή του καπνού. Ε, τα θέματα της ζάχαρης επίσης τα καπνικά προϊόντα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση για τη ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι σαφώς ένα στοιχείο που θέλει να κάνει πιο εύγευστα τα καπνικά προϊόντα και με τον τρόπο αυτό τα κάνει πιο ελκυστικά στους καπνιστές. Κατευθυντήρες γραμμές του ΠΟΕ ΠΟΗ μάλλον, συγγνώμη, λένε ότι πρέπει να απαγορεύσουμε όλες αυτές τις ουσίες που κάνουν πιο ελκυστικά τα τσιγάρα και γι' αυτό υπήρξε φυσικά, όπω ξέρετε, και ο κίνδυνος νομικής προσφυγής εάν υπάρξουν εξαιρέσεις για τη μενθόλη και το ίδιο μπορεί να ισχύσει αν κάνουμε μια εξαίρεση για τη ζάχαρη. Οποιοδήποτε άρωμα ή γευστική ουσία δεν θα πρέπει να επιτραπεί για τα τσιγάρα. Αν θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατότητα να εμποδίσουμε τους καπνιστές και ιδίως τους νέους που ξεκινούν να καπνίσουν, θα ήθελα να έχουμε ένα θετικό κατάλογο και γι' αυτό έχουμε συνυπογράψει με άλλους βουλευτές ένα κατάλογο προσθετικών ουσιών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα καπνικά προϊόντα και πρόκειται μονάχα για αυτές τις προσθετικές ουσίες που έχουν πάρει εκπεφρασμένη έγκριση. Όλες οι άλλες ε, προσθετικές ουσίες θα πρέπει να απαγορεύονται και πρέπει να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Μακάβαν για τις προσπαθίες της και σας ευχαριστώ και σας για την επίοικια που απουσίασε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι σε μια δημοκρατία ο διάλογος θα πρέπει να είναι το αποφασιστικό στοιχείο για την ε, σφυριλάτηση κοινών θεμάτων. Είναι κάπως απώλεια το ότι όλα ορισμένα επιχειρήματα στιγματίζονται και χαρακτηρίζονται ως προεχόμενα από λόμπι και οργανωμένα συμφέροντα. Όπως είπε ο κύριος Φλόρενς. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, μάλλον δεν υπάρχουν επιχειρήματα για ορισμένα σημεία και δεν θα πρέπει να αφήσουμε την ορθολογική συζήτηση και να αφήσουμε τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από τα λόμπι και όλα αυτά. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω με την κυρία Ζόμερ και για όλα αυτά που έλεγξα σε σχέση με τον καφέ επί τη ευκαιρία. Ναι. Ελπίζω ότι δεν θα περιορίσει το χρόνο μου που έχω τρία λεφτά για να μιλήσω. Ας μην μιλήσουμε τώρα για τα θέματα αυτά του καφέ. Συμφωνώ λοιπόν με τη Ρενάτε Ζόμερ και άλλους που είπανε ότι αυτή η οδηγία πηγαίνει πολύ μακριά και είναι πολύ περιοριστική. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε ορισμένες προτάσεις της Κομισιόν για τη συσκευασία. Το να προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες και να είμαστε υπερβολικά περιοριστικοί όπως παγκοσχάρι χάρη στα άρθρα 12 και 13. Γιατί η Κομισιόν τελικά δεν θέλει να αποφασίσει και η ίδια πώς θα είναι πακεταρισμένα τα πακέτα. Αυτό δεν θα αφήσει στη βιομηχανία και στην αγορά κανένα περιθώριο πια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει μια δήλωση στα πλαίσια της ΠΟΗ και έχει αναγνωρίσει ότι οι προειδοποίησεις στα πακέτα μπορούν να εξασφαλίσουν την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Μετά από το 50% θα περάσουμε στο 70% ως ποσοστό κάλυψης των συσκευασιών. Πού ακριβώς είναι η προσθέμενη αξία και ποιο είναι το επιχείρημα το οποίο υποστηρίζει μια τέτοια αντιμετώπιση. Και επίσης για τα προϊόντα, τα τσιγάρα που τα στρίβει κανείς μόνος του η Κομισιόν επιμένει να πολλούνται μόνο σε σακούλες και να απαγορεύσει τα κυλινδρικά δοχεία στα οποία υπάρχουν. Και ποια είναι η λογική, ποια είναι η επιχειρηματολογία που οδηγεί αυτό, γιατί άμα βρίσκονται σε κυλινδρικά δοχεία είναι πιο επικίνδυνα ή πιο αρνητικά από ότι αν είναι σε, σε σακουλάκια. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν αυτή η λογική. Θα ήθελα η Κομισιόν να μα εξηγήσει αν πράγματι υπάρχει κάποια επιχειρηματολογία προ τα θέματα αυτά. Και επίση υπάρχει και μια ακόμα διατύπωση στην πρόταση τη Κομισιόν η οποία είναι ιδιαίτερα περιοριστική. Αν υπάρξει μια ιδέα η οποία θα είναι ε, ενδιαφέρουσα είναι το αυτό που λέει η Κομισιόν ότι δεν πρέπει να μπαίνει τίποτα στην ε, συσκευασία παρά μόνο δηλώσεις που έχουν ένα θετικό χαρακτήρα υπέρ της ανθρώπινης υγείας. Αυτό μου θυμίζει την κομμουνιστική εποχή. Τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί αυτό να καθορίζεται από την Κομισιόν το τι είναι αυτό το οποίο είναι θετικό. Αυτό είναι μια αυθαίρετη αντιμετώπιση από την πλευρά της Κομισιόν, την οποία δεν μπορούμε να δεχτούμε. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η διατύπωση που έχουμε ενώπιόν μας είναι κάτι το οποίο θα μας εκθέσει σε επικρίσεις από την πλευρά των, ε, των ε, πολιτών μας και θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών οι οποίοι θα γίνουν ευρωσκεπτικιστές και θα έχουν μια αρνητική στάση εναντί της Κομισιόν. Ο Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ. Εγώ θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω με εγρήγορση και συνείδηση το θέμα αυτό Βλέπω ότι ο κύριος Φλόρενς ήταν κάπως πιο συγκινησιακός στα θέματα αυτά και όχι κατά ανάγκη ε, ορθολογικός. Ο κύριος Κράμερ είπε για, μια, για τα διοξίδια, για, το, για τις εκπομπές διοξίδιο του άνθρακο σε μια μεγάλη γερμανική εφημερίδα ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια επιτροπή γεμάτη ονειροπόλους. Εμείς έχουμε καταλήξει όμως στο θέμα αυτό σε πολύ καλές ε, λύσεις και, το, και η φιλελεύθερη ομάδα έχει συμμετάσχει σε αυτές τις συμβαστικές λύσεις. Επομένως δεν είναι θετικός ο τρόπος με τον οποίο δήλωσε αυτά τα πράγματα ο κ. Κράμερ. Έρχομαι τώρα στο θέμα. Νομίζω ότι είναι εξισορροπημένη αυτή η πρόταση και αυτό φαίνεται από το μεγάλο αριθμό τροπολογιών που καλύπτουν όλες τις ε, παρατάξεις και πτυχές γιατί ε, για τα πακέτα και τη συσκευασία θα πρέπει να καταλάβει κυρία Μακάβαν ότι είναι υπερβολική η προσπάθεια να έχουμε απλή συσκευασία για τις προσθετικές ουσίες πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Και το πιο σημαντικό ε, είναι οι τροπολογίες για μένα 13.53, 14.54 και 13.55 εμείς με ένα ορισμένο αριθμό συναδέλφων θελήσαμε να τονίσουμε περισσότερο τον κίνδυνο της παθητικής, του παθητικού καπνίσματος, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Όταν εμείς στις Βρυξέλλες, σε οποιαδήποτε από τις χώρες μας, βγαίνουμε στο δρόμο και ε, ρωτάμε τους πολίτες αν ξέρουμε ότι ο καπνί, ε, το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο των πνευμόνων, το ξέρουν οι περισσότεροι από αυτούς. Αλλά το γεγονός ότι οδηγεί σε ευνίδιο θάνατο των νεογνών, ότι μπορεί να προκαλέσει άσθημα και άλλες ε, παθήσεις στα παιδιά και να τις ενισχύσει όταν υπάρχουν, αυτό δεν είναι γνωστό σε όλους και δεν υπάρχει μια τόσο μεγάλη συνείδηση. Πρόκειται λοιπόν για στοιχεία που θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο. Κατανοώ το επιχείρημα της ε, ελευθερίας. Ο καθένας μπορεί να αποφασίσει αν κάνει κακό στον εαυτό του ή όχι, αλλά όχι για τα παιδιά. Δεν μπορεί να αποφασίζει ο ίδιος τι θα κάνει για τα παιδιά του. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτές οι τροπολογίες θα πρέπει να τύχουν υποστήριξη. Η Κομισιόν λέει ότι αυτά τα θέματα δεν έχουν καμία σχέση με το νομοθέτημα αυτό, αλλά πρέπει να ρυθμιστούν σε επίπεδο επιτροπολογίας. Κύρια Κομισιόν, εμείς έχουμε όμως ένα ρόλο συναπόφασης σε αυτό το νομοθέτημα. και δεν θέλουμε να συζητούμε όλα αυτά τα πράγματα επί εβδομάδες και μετά η Κομισιόν έχει τον τελικό λόγο μέχρι τις επιτροπολογίες. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να περιορίσουμε ιδιαίτερα το τμήμα της πρότασης αυτής που υπόκειται στην επιτροπολογία και ζητώ να υποστηρίξετε τις τροπολογίες μας. Ο κύριος Μπάολο Μπαρτολότσι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την εργασία που έχει κάνει. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μαζί με άλλους Ιταλούς συναδέλφους που είναι μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος έχουμε υποβάλει διάφορες τροπολογίες πολύ άριθμες στο κείμενο αυτό και όλες αντικατοπτρίζουν τις ε, σοβαρές μας ανησυχίες σε σχέση με αυτές τις ε, προτάσεις που αν υιοθετηθούν και εγκριθούν θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, την ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά και άρα ε, και συνέπειες για την ε, απασχόληση και άρα και για τους πολίτες και δεν φαίνεται να επιτυχάνουν με, επιτυχε... με τους στόχους της δημόσιας υγείας. Ε, και μάλιστα έχουμε σοβαρές αμφιβολίες. Αναφέρομαι στην ίδια τη βάση, τη νομική βάση που έχει επιλέξει η Κομισιόν και που σχέζεται, σχετίζεται με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών και τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Οι στόχοι αυτοί αντικατοπτρίζονται στην πρόταση κειμένου και αντικατοπτρίζεται η ίδια ομόφωνη γνώμη που έχουν εκφράσει πολλά εθνικά κοινοβούλια, όπως για παράδειγμα και οι αρμόδιες επιτροπές της, ε, του Ιταλικού Κοινοβουλίου και της Γερουσίας και που, ε, που έλαβαν αντική θέση όσον αφορά την επικουρικότητα για τη συγκεκριμένη πρόταση οδηγία. Τώρα, οι απαγορεύσεις που προβλέπονται, ας πούμε, ε, από την απαγόρευση των τσιγάρων ε, slim και όλες τις άλλες, αναφέρονται στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, θα, και, και, και διακινδυνεύουν μια εναρμόνιση ομοιόμορφη. Ο ίδιος προβληματισμός όσον αφορά δηλαδή τα απλά πακέτα ή την ομοιομορφία των πακέτων. Εδώ μπορεί να επιδεινωθεί ο ρόλος του ελέγχου και επίσης το θέμα των ε, φόρων, ε, της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας, ενημέρωσης προς καταναλωτές, αλλά και της συμφωνίας TRIPS Ανάλογες είναι οι ανησυχίες για τα μέτρα που καθιστούν πιο δύσκολη την πρόσβαση στα προϊόντα και που παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο τα προϊόντα, δηλαδή μικρότερο κίνδυνο για τα οποία δεν υπάρχει ad νομικό πλαίσιο και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα τα οποία, για τα οποία ήδη υπόθηκαν πολλά. Τελευταίες ανησυχίες τέλος για τις διάφορες διατάξεις που δίνουν αρμοδιότητες στην Κομισιόν ακόμα και σε πολύ σημαντικά στοιχεία. Τέτοιες ε, αρμοδιότητε, κανονικά τα έπρεπε να, είναι περιορισμένες και να κατα... τελικά τα μέτρα αυτά που προτείνονται στην ουσία θα τους αφιβολία το αρμοδιότητες των ε, κρατών μελών. Όλα αυτά, ε, όλες αυτές οι ανησυχίες αντικατοπτρίζονται στις τροπολογίες που υποβάλαμε και που θέλουν να ε, ε, παρεμποδίσουν τη λήψη αποφάσεων που είναι αντίθετες ε, όχι μόνο με τους στόχους που υποτίθεται ότι έχει αυτή η πρόταση, αλλά θα ενθάρρυναν και μια μεγάλη αύξηση του λαθρεμπορίου. Παράνημες πωλήσει λοιπόν ε, θα αυξάνονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παραμένω ωστόσο πεπισμένος ότι πιο σχετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη μέτρα για τον περιορισμό του καπνού θα ήταν αν μπορούσαμε να ε, υποβάλουμε προτάσεις ώστε να δεσμευθούν η παραγωγή και τα θεσμικά όργανα, ε, ώστε να επενδύσουν σε σε πρόληψης και ενημέρωσης, ε, όπου θα συμμετέχουν και θα ενημερώνονται οι πολίτες, οι καταναλωτές και κυρίως οι νέοι, καθώς και οι έγκυες γυναίκες. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με πολλά που είπε η Ματίνα Συγχαίρω την Ιρλανδική Προεδρία για τη στάση της. Θαυμάσια ναι. Με λυπεί όμως ε, κάπως συζήτηση. Ακούω ορισμένους να παρομοιάζουν το κάπνισμα με το, με το καφέ. Πέφτει το επίπεδο της συζήτησης. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε το κάπνισμα. Όχι, δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε το δικαίωμα επιλογής. Αλλά δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τη σημασία για τη δημόσια υγεία που έχει ε, το θέμα αυτό. Ένας από τους δύο καπνιστές θα πεθάνει επειδή καπνίζει. Τεράστιο κόστος ε, για τους προπολογισμού υγείας, τεράστιο ανθρώπινο κόστος κυρίως. Δεν είναι μικρό θεματάκι. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να το επιβάζουμε έτσι, να το εξευτελίζουμε έτσι. Έχω υποβάλει πολλές τροπολογίες με συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες. Δεν θα μπω σε αυτές τις τροπολογίες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ωστόσο. Πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως οποιοδήποτε άλλο προϊόν υποκατάστασης του καπνίσματος. Κανείς δεν θα μου αλλάξει τη γνώμη γι' αυτό. Αλλά κάτι συγκεκριμένο. Ε, πώς ε, εμφανίζονται τα προϊόντα καπνού στα σημεία πώλησης. Μια σειρά από κράτη-μέλη εφαρμόζουν απαγορεύσεις στην επίδειξη των προϊόντων καπνού στην, ε, στα σημεία πώλησης και έχει αποδειχθεί ότι έτσι ε, περιορίζεται το ενδεχόμενο να αρχίσουν να καπνίζουν οι άνθρωποι και ιδίω οι νέοι. Στη Νέα Ζηλανδία αποδείχθηκε ότι αν υπάρχει επίδειξη των προϊόντων καπνού τριπλασιάζεται το ενδεχόμενο να αρχίσουν να καπνίζουν οι νέοι. Αυτό είναι σαν διαφημιστικές ε, ταμπέλες για τις ε, εταιρείες ε, τσιγάρων. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να συνεχίσουν να κρύβονται τα τσιγάρα. Ορισμένοι θα πούνε ότι δεν είναι ενωσιακή αρμοδιότητα, αλλά οι βιομηχανίες τσιγαρέτων, τσιγαρέτων ε, κάνουν μηνύσεις ε, όπως στην Νορβηγία το 2011 κατά των κυβερνήσεων λέγοντας ότι προκαλούν στρέβλο στην αγορά. Έχω ακούσει μια φήμη ότι υπήρχε αυτή η απαγόρευση στην αρχική πρόταση της Κομισιόν και βγήκε τελευταία στιγμή. Λυπάμαι γι' αυτό. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αυτό το μέτρο για να εμποδίσουμε τους νέους να αρχίσουν να καπνίζουν και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για να σώσουμε την επόμενη γενιά από αυτή την ασθένεια, τους θανάτου και τις αναπηρίες που προκαλεί το κάπνισμα. Ηρέλιο Ροντρίγκεθ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι φιλόδοξη πρόταση δεν θα κάνουμε αυτή την τροποποίηση της προηγούμενης οδηγίας για να οπισθοχωρήσουμε. Βλέπω όμως ότι έχει υπάρξει τρομερή πίεση από τα λόμπι στην Ισπανία για παράδειγμα που παράγεται καπνός, καλλιεργείται καπνός όπου ακούσαμε ε, πολλά πράγματα που δεν ισχύουν και όμως γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες που προσπαθούν να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ των θέσεων που θέλουν πλήρη απαγόρευση και των θέσεων που θέλουν να διατηρηθεί η κερδοφορία του κλάδου. Για παράδειγμα, θα πρέπει να διατηρηθεί η εξαίρεση για τα πουρα. Διότι όπως ξέρετε κανένας δεν ξεκινάει να καπνίζει καπνίζοντας πουρα και ιδίως οι νέοι. Γιατί είναι και ακριβά και καπνίζονται αργά. Πιστεύω το 10% είναι καλό, αλλά για να δούμε ποιες είναι οι χώρες που καμνίζουν πιο πολύ, θα δούμε ότι είναι σημαντικές αυτές οι χώρες. Πρέπει να καταργήσουμε τα πρόσθετα. Όποιος θέλει να καπνίσει καπνό, καπνίζει καπνό, δεν καπνίζει φράουλες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν πάρα πολλά πρόσθετα. ούτως ή άλλως κατά την κατεργασία του φύλου του καπνού μειώνεται ένα ποσοστό από τη ζάχαρη. Όπως για παράδειγμα κατά την ε, κατεργασία της, ε, ε, του χυμού του, στο πορτοκάλι χάνουμε ένα ποσοστό καπνού. Άρα το να προσθέσουμε κάποια ζάχαρη δεν είναι τόσο τεχνητό. Πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε συμφωνίες χωρίς να χάσουμε από ε, το νου μας το στόχο. Ο στόχος είναι να μην αρχίσουν να καπνίζουν οι νέοι και να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό η οδηγία αυτή ε, υπογράφεται από ε, τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για την υγεία και το συζητάμε εδώ στην Επιτροπή που είναι αρμόδια για την υγεία. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε στον κλάδο σε όλους. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε στο κέντρο της προσοχής μας τη δημόσια υγεία χωρίς όμως να γίνουμε τόσο απόλυτοι που να ε, προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάτι ανέφικτο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Δελάνια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, όπως και πολλοί άλλοι, αλλά όλοι, όχι όλοι που άκουσα, δικό μου στόχος θα ήταν η μηχανία να μην αποκτήσει νέους καταναλωτές ή χρήστες και ότι αυτοί που υπάρχουν δεν θα βλάψουν τους υπόλοιπους. Και είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε από αυτή την άποψη ότι από τότε που απαγορεύτηκε το κάπνο στο Βέλγιο σε όλα τα εστιατόρια και μπαρ, ο, ο αριθμός των ευνηδίων των πρόωρων γεννήσεων έχει μειωθεί πολύ σημαντικά. Είναι ένα, μια από τις παρενέργειες του καπνίσματος στα βρέφη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ακόμα ένα θέμα στα τρία λεπτά που έχω, ότι ήδη το, η σύμβαση πλαίσιο για το καπνό λέει πως ε, τα συμβαλόμενα μέρη θα πρέπει να απαγορεύσουν τη χρήση προϊόντων που στόχο έχουν τα παιδιά, δηλαδή τα παιχνίδια και εκείνες τη σοκολατένια τσιγάρα, ε, Λίντα, που και εγώ πήρα πριν από τα Χριστούγεννα την γιορτή του Αγίου Νικολάου. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι δίνεις τη τσιγάρα στα παιδιά γιατί μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ε, για να μιμηθούν ε, τους καπνιστές. Ε, δεν έχουν ακόμα όμως απαραλευθεί παρόλα αυτά. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν πιο προηγμένα παιχνίδια από τις σοκολάτες και τα, οι τσίχλες που ξέραμε εμείς. Υπάρχει το στυλό ναργιλές που μιμείται τον ναργιλέ και έχει και γεύση. Δεν ξέρουμε καταρχήν αυτή η γεύση τι προκαλεί στην υγεία, δεν υπάρχει σχετική έρευνα και έπειτα είναι πολύ ελκυστικά για τα μικρά παιδιά γιατί είναι κάτι γυαλιστερά, πράσινα, ροζ, ε, στυλό ε, έχουν και ένα φωτάκι στην άκρη τους και μάλιστα όταν σε εκείνο το φωτάκι ανάβει, κόκκινο γίνεται. Ε, φανταστικό για τα παιδιά. Και τα παιδιά έχουν πρόσβαση ε, σε όλα αυτά. Κατά τη γνώμη μου, ένας βασικός δηλαδή λήθος για την, την βιομηχανία για να αρχίζουν τα παιδιά να καπνίζουν. Και αυτά δεν καλύπτονται ούτε από αυτήν την οδηγία. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε αυτά όλα να απαγορευτούν, όπως και τα τσοκολατένια τσιγαράκια για τα παιδιά είναι δύσκολο να πλαισιώσει κανείς νομικά, να βρει μια διατύπωση και να απαγορεύσει αυτά τα προϊόντα. Εγώ προσπάθησα να το κάνω μέσω μιας κατηγορίας ε, προϊόντων μίμησης καπνού ή καπνίσματος. Σε πάση περιπτώσει δεν με ενδιαφέρει πώς ε, θα το διατυπώσουμε από τη στιγμή που θα γίνει. Και τέλος για τις κατεξοδότητες συμπράξεις, παρακαλώ να γνωρίζετε πως δεν είναι μόνο το δικό μας σώμα που θα πρέπει να ανησυχεί για την προσπάθεια της ε, Κομισιόν να ελκύσει όλη την αρμοδιότητα για να τροποποιήσει αυτήν την οδηγία στον εαυτό τη. Δεν, να δε στην Κομισιόν δεν είναι άμεσα εκλεγόμενο σώμα, αλλά και πολλά εθνικά κοινοβούλια ε, θα αν, αν δώσουμε σε αυτή, στην Κομισιόν αυτή την υπερβολική εξουσία, την υπερβολική αρμοδιότητα για να κάνει τι επόμενε μερικέ ή πλήρε αναθεωρήσει μέσω κατεξοδότηση πράξεων θα, και τα εθνικά κοινοβούλια ανησυχούν ανησυχούν γι' αυτό. Ξέρω πως ανησυχεί σίγουρα το Ολλανδικό Κοινοβούλιο και στηρίζω τη Λίντα εδώ που λέει ότι θα πρέπει όντως να περιορίσουμε τις φιλοδοξίες της Κομισιόν σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πρώτα τη Λίντα για αυτά που είπε για το σνούς, ότι πρέπει να υπάρξει δυνατότητα επιλογής. Ή πρέπει να το επιτρέψουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να σεβαστούμε την ιστορική παράδοση όπως καταγράφεται και στη συνθήκη ένταξης των, της Σουηδίας και να εξαιρεθεί από αυτήν την ρύθμιση. Δεν είναι επαρκές να το αφήσουμε κατά μέρος. Πρέπει να δώσουμε μία λύση. Γιατί αυτά που έχουμε τώρα αλλάζουν την τωρινή κατάσταση του status quo. Γιατί λέμε ότι το ρυθμίζουμε το θέμα αυτό μόνο στη Σουηδία και το απαγορεύουμε σε όλη την εσωτερική αγορά. Ξέρω ότι έχετε βαρεθεί αυτό το θέμα. Αλλά αν θέλουμε να επιτρέψουμε τα σιγάρα και να απαγορεύσουμε το σνούς και να το ρυθμίσουμε μονάχα στη Σουηδία, είναι σαν να λέμε ότι απαγορεύουμε τη βότκα και ρυθμίζουμε τα θέματα του ίνου μόνο στη Γαλλία. Αυτό θα ενοχλούσε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ, μεταξύ των δύο επιλογών, Θέλω να επιχειρηματολογήσω υπέρ της ε, έγκρισης του σνούς σε όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη προστασία ή απαγόρευση. Αυτά που ελέγχθηκαν προηγουμένως για τα τσιγάρα είναι σωστά. Είναι παράλογο να έχουμε για ορισμένα προϊόντα λιγότερη προσβασιμότητα από ό,τι στα τσιγάρα, για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα παραδείγματος το σνους είναι λιγότερο επικίνδυνο και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία της Σουηδίας. Το πρόβλημα του καπνού είναι όταν καίγεται ο καπνός. Τότε είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο. Το σνούς δεν καίγεται, επομένω δεν έχει τόσο κίνδυνο για την υγεία. Όλα τα άλλα είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Άμα κάθεστε και αναπνέετε από τις εξατμίσεις των αυτοκίνητων και αυτό είναι τρομερά επικίνδυνο και μπορεί να σας σκοτώσει. Το λοιπόν είναι ένας τρόπος να χρησιμοποιείται κανείς τον καπνό χωρίς να έχει όλα αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα από την καύση. Καταλαβαίνω. Ότι το να το εγκρίνουμε, το να το επιτρέψουμε δεν είναι ίσως η σωστότερη γραμμή, αλλά ούτε είναι και να το απαγορεύσουμε απόλυτα. Όπως είπε και η φίλη μας από την ε, συντηρητική ομάδα, δεν είναι μονάχα ένα θέμα που αφορά μόνο τη Σουηδία και στη Δανία υπάρχει μεγάλη διαμάχη για το σνούς. Και στην Νορβηγία που είναι μέρος της ΕΖΕΣ και εκεί υπάρχει επιρροή για τα θέματα αυτά. Είναι κάτι το πολιτιστικό. Νομίζω λοιπόν ότι η μόνη λογική λύση είναι να πούμε ότι τα κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να διατηρήσουν το σνούς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το διατηρήσουν όπως έχουν τώρα. Κάπου αυτό πρέπει να γραφτεί στο κείμενο λοιπόν, σαν συμβιβαστική λύση. Αλλά το να παραγωνίσουμε το θέμα αυτό και να μην πούμε τίποτα, αυτό δεν είναι λύση. Θα πρέπει να δεχτούμε τουλάχιστον κάποιες τροπολογίες για να διατηρηθεί το σνούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Έντιδε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Λίντα Μακέβν για το πολύ δύσκολο έργο που χρειάστηκε να φέρει σε πέρας για αυτό το τόσο αμφιλεγόμενο θέμα και το έκανε με μεγάλη σοβαρότητα. Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι ένας στόχος που συμμεριζόμαστε όλοι και που θέλουμε να τον προωθήσουμε. Είναι αποδεδειγμένο ότι ο καπνός βλάπτει την υγεία και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι καπνιστές και ιδίως οι νέοι να έχουν μια επίγνωση των κινδύνων που έχουν ενώπιόν τους. Αλλά κυρίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ανάγκη να είμαστε λογικοί. Σε ό,τι αφορά παραγωγή χάρη τις καπνοβιομηχανίες, εγώ θεωρώ ότι έχουν δίκιο όταν λένε για τον κίνδυνο αύξηση της λαθρεμπορίας τσιγάρων και της παραποίησης των τσιγάρων. Είναι απαραίτητο να αποφύγουμε λοιπόν την αύξηση της παραποίησης και του λαθρεμπορίου. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, όπως ελέγχθη, στην Πορτογαλία κάθε μορφή διαφήμισης για τα καμνικά προϊόντα απαγορεύεται. Οποιαδήποτε μορφή έμεση, άμεση, απαγορεύεται. Εγώ έχω παρουσιάσει για το, την παράγραφο 8 μία τροπολογία και θα ήθελα η Λίντα να με υποστηρίξει εδώ. Στην τροπολογία παρουσίασα μαζί με άλλους Πορτογάλους συναδέλφους και που έχει να κάνει με τα θέματα συ... συσκευασίας. Έχουμε ε, ένα πλάτος 53 χιλιοστών μονάχα και ένα μεταβλητό ύψος των πακέτων. Μικρότερα πακέτα από άλλες περιοχές και ιδίως στις αυτόνομες περιοχές της ε, Μαδέρας και των Αζωρών θα μια αλλαγή στις προδιαγραφές για την έκταση των προειδοποίησεων θα έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, αντίκτυπο σε αυτές τις περιοχές όπου η καπνοβιομηχανία έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις και για μια τέτοια αλλαγή θα είχε πολύ αρνητικό ε, αποτέλεσμα, θα οδηγούσε σε μια αύξηση της ανεργίας που είναι ήδη πολύ υψηλή στην περιοχή αυτή, στις περιοχές αυτές. Αυτό λοιπόν δεν έχει καμία επίπτωση στην ε, ανθρώπινη υγεία, το να είναι πιο ε, βραχία τα τσιγάρα ή να είναι πιο μικρές οι συσκευασίες, αυτό δεν αλλάζει την ε, θέληση των καπνιστών να καπνίζουν ή να σταματήσουν το κάπνισμα. Και για το ίδιο αυτό λόγο είμαστε εναντίον της ε, πρότασης από τους φιλελεύθερους να αυξηθούν οι διαστάσεις των ε, συσκευασιών και των προειδοποίησεων. Αυτό θα οδηγήσει και σε προβλήματα για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν είναι ακριβώς αυτό το μείγμα μας αφορά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το θέμα της συσκευασία, αλλά είναι το θέμα της δημοσίας υγείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Γκαρτίνη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά πράγματα έχουν ήδη υποθεί και έχω την εντύπωση πως εν γέννη θα μπορούσαμε να πούμε πως όλοι είμαστε στην ίδια γραμμή όταν λέμε πως συμφωνούμε με το γεγονός ότι ο καπνός βλάπτει και άρα πρέπει να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η χρήση του καπνού. Επίσης συμφωνούμε όταν λέμε ότι η προτεραιότητα είναι να προστατευτούν οι νέοι, να μην ε, διευκολύνουμε και να παγορεύσουμε μάλλον να υπάρξουν νέα νέοι καταναλωτές και ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από το υπαθητικό κάπνισμα, όπως είπε πολύ ωραία ο συνάδελφος Λίζε. Ωστόσο, όλα αυτά γίνονται και γίνονται με πιο αποτελεσματικά μέσα. Δεν συμφωνούμε για τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την επιτευξή των στόχων. Η πρώτη φορά, για παράδειγμα, που η Ευρώπη, που συνήθως προσπαθεί να θεσπίσει εναρμονισμένους κανόνες για θέματα σήμανσης των προϊόντων, αυτή τη φορά αφιερώνεται και στο μορφή, στο σχεδιασμό του πακέτου του κανόνες που βασικά είναι πιο εμπορικοί από ότι η προστασία της υγείας. Εγώ είμαι Ιταλίδα. Δεν πιστεύω πως η Ιταλία όπως άκουσα από αλλού ε, έχει αμφίσιμη στάση. Η Ιταλία εδώ και χρόνια αγωνίζεται κατά του καπνού. Μάλιστα, ε, μελέτες ε, της γερουσίας της Ιταλίας μας λένε ότι από το 2003 μέχρι το 2012 το ποσοστό των καπνιστών από 27,6% πέρασε στο 20,3%. Ε, ε, δηλαδή ένα πολύ χαμηλότερο ποσοστό και με στρατηγικές πολύ διαφορετικές από αυτές που τώρα θέλουν να μας υποδείξει Κομισιόν. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Εστρέλα που μόλις μίλησε. Δεν βλέπω τι διαφορά μπορεί να έχει για έναν καπνιστή το να έχει ένα τσιγάρο πιο μακρύ, πιο κοντό, πιο χοντρό ή συσκευασμένο σε διαφορετικό τρόπο. Εγώ περισσότερο πιστεύω στους χώρους πώλησης, στην εκπαίδευση των παιδιών που θα πρέπει από τα σχολεία να γνωρίζουν τους κινδύνους ε, και είναι μάλιστα και ένα πράγμα που κάναμε. Έχουμε και Ελβετούς ερευνητέ που είπαν που, ε, πήραν καπνιστές, δηλαδή που είναι εξαρτημένοι από τη χρήση ενός προϊόντος, να δεν το βρούνε σε μια αγορά θα πάνε να το βρουν αλλού. Τα στοιχεία μας λένε ότι όχι τόσο το λαθρεμπόριο του τσιγάρων αλλά η παραποίηση τσιγάρων είναι ε, σαφώς αύξηση. Ε, ε, για ένα λόγο γιατί αυτό οδηγεί η κρίση τους πιο ευάλωτους και τους πιο φτωχούς να στραφούν προς αυτό το είδος εμπόριο. Και έπειτα τι ξέρουμε για αυτά τα τόσο επικίνδυνα τσιγάρα, τα παραποιημένη. Απολιγμένα τσιγάρα, σε μολυσμένα τσιγάρα, ακόμα και κομμάτια πλαστικού μέσα μέσα σε αυτά τα τσιγάρα, τα παραποιημένα. Δηλαδή, εκτιθέμεθα εκτιθέμεθα όχι μόνο σε ένα κίνδυνο μεγαλύτερο για την υγεία αργότερα, αν δεν σταματήσουμε αυτή την αύξηση της παραποίησης που το απλό πακέτο θα διευκόλυνε, ε, όπως δείχνουν οι μελέτες, αλλά θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πολύ σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας. Φανταστείτε τι θα γίνει άμα υπάρξουν δηλητηριάσεις από υλικά άγνωστα, γιατί στα παραπημένα τσιγάρα δεν ξέρουμε καν τι βάζουν μέσα. Αυτή είναι, εδώ υπάρχει διάγνωση μεμονωμένων περιπτώσεων δηλητηρίασης αλλά και πιο μακροπρόθεσμων, μακροχρόνιων ασθενειών. Και κλείνω γιατί πέρασε ο χρόνος μου και για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ανησυχούμε πολύ αλλά εκτείνοντας στο τμήμα των προϊόντων μειωμένου κινδύνου νέας γενεάς πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ευρύτερη, ένα ευρύτερο προβληματισμό γιατί έτσι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμποδίσει τα κρατημέλη να εισάγουν μια πολιτική περιορισμού των κινδύνων που προκύπτουν από τα προϊόντα καπνού. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε και ευχαριστώ με την ευκαιρία και την συγκήτρια που κάνει το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε εδώ έκλεισε ο κατάλογος των ομιλητών είναι μία από τις μεγαλύτερες νομοθετικές ε, διαδικασίες που έχει επιτελέσει η Επιτροπή μας και ιδιαίτερα επίμαχη. Είναι γεγονός ότι ε, πεθαίνουν 700.000 άτομα το χρόνο μέσω του καπνίσματος στην Ένωση. Εάν ε, κάνουμε τον υπολογισμό ανακράτος μέλος, όπως έκανε ο Καρλ Χάινς Φλόρεντς, εάν κάθε μέρα έπεφτε ένα αεροπλάνο σε κάθε κράτος μέλος, σε τρεις μέρες θα είχε απαγορευτεί ε, η ενέργεια κυκλοφορία. Όμως δεν έχουμε επιβάλει τέτοια απαγορεύση για το καπνό. Αυτό είναι το δίλημα που έχουμε μπροστά μας. Βέβαια είναι δύσκολο για έναν εξιντάρι ε, που καπνίζει ε, δεκαετίες να σταματήσει να καπνίζει επειδή θα του το απαγορεύσουμε. Βεβαίως ε, έχουμε τώρα αυτό το νομοθέτημα μπροστά μας και στόχος είναι να μην αρχίσουν οι νέοι να καπνίζουν, να μην αποκτήσουν οι επόμενες γενιές αυτήν την εξάρτηση. Αυτός είναι ο στόχος αυτού του νομοθετήματος. Στην περιοχή μου υπάρχει μια παροιμία. Πρέπει η εκκλησία να είναι στη μέση του χωριού, δηλαδή να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Θα ήταν σκόπιμο λοιπόν να επιχειρήσουμε να το καταλάβουμε αυτό, να προωθήσουμε τη δημόσια υγεία, να μην αρχίσουν να καπνίζουν πολύ, αλλά και για τα καινοφανή προϊόντα. Κάναμε μία συνεδρίαση γι' αυτό, ένα σεμινάριο. Δεν ε, με ικανοποίησαν τα συμπεράσματα του σεμιναρίου αυτού για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, γιατί έχουν ε, εισαχθεί αυτές οι οριακές τιμές που στην ουσία απαγορεύουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο και μπορεί κανείς να το αγοράσει μόνο στα ε, ε, φαρμακεία. Εντάξει, εμένα μπορεί να μου αρέσουν, αλλά όσοι θέλουν να θα κόψουν το κάμψιμα και να συνεχίσουν να ε, προσλαμβάνουν νοικοτήνη, μπορούν να το αξιοποιήσουν. Αλλά για το θέμα αυτό θα πρέπει να το συζητήσουν οι συγητές, οι συνεισηγητές και στο τέλος αυτής της διαδικασίας η Λίντα Μακάβαν θα πρέπει να εξετάσει αυτές τις 1300 ε, τροπολογίες. Ελπίζω βέβαια να μειωθούν. Αυτό το νομοθέτημα θα πρέπει να το αποφασίσουμε μέχρι τις ευρωεκλογέ. Αυτή πρέπει να είναι η πρόθεσή μας. Πιέσαμε την Κομισιόν να μας υποβάλει όσο το δυνατόν νωρίτερα αυτό το κείμενο. Ξέρουμε τι δυσχέρειες είχε η Κομισιόν, άλλαξε και ο Επίτροπος. Αλλά η Επιτροπή λίγο πριν τα Χριστούγεννα μας υπέβαλε την πρόταση ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι ε, περιμέναμε και αυτό μας κανοποίησε. Πρέπει λοιπόν και εμείς να βιαστούμε να καταλήξουμε σε κάτι θετικό με βασική προϋπόθεση να κρατήσουμε την εκκλησία στη μέση του χωριού. Ε, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να είναι στρογγυλέ ή τετράγωνε οι συσκευασίε. Εντάξει, αλλά έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην εισηγήτρια ότι θα τα καταφέρει. Και πριν δώσω το λόγο για το κλείσιμο στην ε, εισηγήτρια, ε, η Κομισιόν παρακαλώ, ε, ετέθησαν πολλά ερωτήματα, πήραμε τον χρόνο που χρειαζόταν, τον αναγκαίο για να συζητήσουμε αυτό το θέμα και παρακαλώ να απαντήσετε στα ερωτήματα των συναδέλφων. Και μετά η εισηγήτρια. Ευχαριστώ ναι. πρόεδρε. Πρώτον, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους κοιόδης και τα μέλη για τα σχόλια, ερωτήσεις και τροπολογίες. Να ε, επαναλάβω την αιτιολόγηση της πρόταση της Επιτροπής. Πρώτον, για τη ρύθμιση των συστατικών. Είμαστε υπέρ της απαγόρευσης ε, όλων των, των ε, προσθετικών που έχουν ισχυρή μη βανίλιας ή φράουλας, γιατί αυτά ε, καθιστούν αυτά τα προϊόντα πιο ελκυστικά για τους νέους και άρα είναι πιο εύκολο να αρχίσουν να καπνίζουν. Βλέπουμε πολλές τέτοιες γεύσεις, βανίλια, κεράσι, τσοκολάτα, καινοφανή προϊόντα, καψούλες με, την, ε, με μεντόλι και αυξάνεται σε, σε πολλά κράτη-μέλη ε, το ποσοστό αγοράς των τσιγάρων με μεντόλ και έτσι μπορεί να περάσει κανείς από, απλή, ε, από το απλό να δοκιμάζει σε κανονικό κάπνισμα. Βλέπουμε ότι και σε άλλες ε, ομάδες ηλικία ε, βοηθάει να αρχίσει κανείς να καπνίζει. Και ε, αυτές οι θετικές γεύσεις κάνουν πιο δύσκολο να καταλάβεις ότι είναι επιβλαβές το κάπνισμα. Συσκευασία και ετικέτες. Οι μελέτες καταδεικνύουν ότι οι μεγαλύτερες προειδοποίησεις, μεγαλύτερες εικόνες είναι θετικές, μειώνουν την κατανάλωση. Το ανάφερε και η συγγήτρια. Άρα γι' αυτό προτείνουμε το 75% κάλυψης. Νομίζουμε ότι είναι ισορροπημένη αυτή η πρόταση. Και όπως υπόθηκε, στο Βέλγιο για παράδειγμα, που πρέπει ήδη να χρησιμοποιεί κανείς τρεις γλώσσες για τις προειδοποιήσεις, ήδη οι τρεις προειδοποιήσεις καλύπτουν 65%. Και η εμπειρία από τον Καναδά. Έχουμε στοιχεία ότι το 75% βοηθάει. Έχουμε λοιπόν ε, επιχειρήματα για το 75%. Δεν είναι τυχαίο ποσοστό. Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα τώρα. Να διευκρινίσω την άποψή μας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αποτελεσματικά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Είναι ασφαλή προϊόντα για να κόψει κανείς το κάπνισμα. Θέλουμε ασφαλή προϊόντα και αποτελεσματικά και καλής ποιότητας προϊόντα για να κόψει κανείς το κάπνισμα. Τρία ερωτήματα λοιπόν τίθενται. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλή και σέβονται τις σωστές διαδικασίες παραγωγής. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό βοήθειας ε, για να σταματήσουν οι καταναλωτές το κάπνισμα και πώς θα εμποδίσουμε να αξιοποιηθούν αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα να οδηγήσουν αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στο να συνηθίσουν το κάπνισμα και την πρόσληψη νοικοτήνης οι νέοι. Τα μελετήσαμε όλα αυτά και θεωρήσαμε ότι τα τσιγάρα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που έχουν νοικοτήνη πάνω από ένα κατόφλι πρέπει να θεωρηθούν φαρμακευτικά προϊόντα. Εξετάσαμε και το δεχόμενο ενό ειδικού καθεστώτος αλλά λόγω λοιπόν των ερωτημάτων που θέσαμε και των μελετών που λάβαμε από τις μελέτες που παραγγείλαμε, πιστεύουμε κατηγορηματικά ότι είναι σκόπιμη η πρότασή μας και θα έχει αποτελέσματα. Τέλος, για την ανακοίνωση για τη λαθρεμπορία. Στις 5 Ιουνίου θα ε, υιοθετήσουμε μία ανακοίνωση και ε, ένα σχέδιο δράσης για τη λανθρεμπορία σιγαρέτων. Θα την εισαγάγει ο Επίτροπος Σεμέτα για τις κατεξιοδότες πράξεις. Παρακολουθούμε τις επιστημονικές εξελίξεις για τον τομέα αυτό Υπάρχουν μια σειρά από τεχνικά θέματα που πρέπει να ρυθμίζονται μέσω τέτοιων πράξεων. Διότι είναι περιορισμένη η δυνατότητα που έχει να χρησιμοποιήσει η Κομισιόν αυτές τις ε, εξελίξεις στην επιστημονική γνώση. Υπάρχει ε, κάποια κινητικότητα και στο Συμβούλιο για να ρυθμιστεί καλύτερα ο τρόπος χρήσης των κατεξοδότηση ε, πράξεων, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε επαρκή ευελιξία στην Κομισιόν για να μπορεί να προσαρμόζει τις ρυθμίσεις στην εξέλιξη ε, της έρευνας. Λέμε ότι στόχος μας είναι μείωση 2% στην κατανάλωση. Ορισμένοι λένε ότι είναι περιορισμένος αυτός ο στόχος. Αλλά το 2% είναι 2,5 εκατομμύρια. Δεν θα έχει λοιπόν τέτοια τεράστια επίπτωση στον κλάδο, αλλά θα έχει τεράστια επίπτωση στη δημόσια υγεία. Ε, η κυρία Βίμερ ίσως θα μπορούσε να εξηγήσει το θετικό κατάλογο ουσιών και την ε, προστίκη ζάχαρης. Για τον θετικό κατάλογο θέλω να αναφέρω ότι η Κομισιόν έχει εξετάσει το θέμα αυτό, έχει αναλύσει τις δυνατότητες και για διάφορους λόγους. Σε αυτή τη φάση είχαμε αποφασίσει να μην προτείνουμε ένα θετικό κατάλογο. Καταρχήν γιατί είναι πολύπλοκος ο χώρος, υπάρχουν χιλιάδες προσθετικές ουσίες σε χρήση και πολλές άλλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Είναι πολύ εύκολο να αντικατασταθεί η μία από την άλλη και είναι πολύ δύσκολο σε επίπεδο ρυθμιστικού ελέγχου να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Επίσης ένας θετικός κατάλογος θα έδινε τη λανθασμένη εντύπωση ότι αυτές οι προσθετικές ουσίες κάνουν πιο ασφαλές το, προϊόντο, το προϊόν και καλύτερο προς τους καταναλωτές. Αυτή είναι μια εντύπωση που δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε γιατί τα προϊόντα του καπνού πάντα είναι βλαβερά. Επίσης, αν ακολουθήσουμε την οδό του θετικού καταλόγου, θα πρέπει να αναπτύξουμε ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια και κανείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ακριβώς τι κριτήρια θα έπρεπε να είναι αυτά να εστιάσουμε στα θέματα του εθισμού, της τοξικότητος, της ελκυστικότητος, της ε, διευκόνσης της εισπνοής του καπνού. Όλα αυτά είναι πολύ, πολύπλοκα σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο. Αν λοιπόν πάρουμε στα σοβαρά αυτό τον θετικό κατάλογο θα καταλήγαμε πολύ πιθανώς σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπος τους καπνοκαλλιεργητές στην Ευρώπη. Γι' αυτό η Κομισιόν ακολούθησε μια πιο εξισορροπημένη προσέγγιση στον τομέα αυτό. Επίσης, θα ήθελα να σας επισημάνω το γεγονός ότι η διαχείριση ενός τέτοιου καταλόγου θα είχε σημαντικό διοικητικό άχθος και θα απαιτούσε πολλούς ανθρώπινους πόρους. Γι' αυτό η Κομισιόν δεν έχει προτείνει ένα θετικό κατάλογο. Θέλω επίσης να σταθώ στο θέμα της τυποποίησης των συσκευασιών και θέλω να σας κάνω σαφές ότι η Κομισιόν δεν προτείνει την ε, τυποποίηση όλων των προϊόντων, των συσκευασιών. Για προϊόντα εκτός των τσιγάρων υπάρχει ένα ευρύτατο φάσμα δυνατοτήτων συσκευασίας. Μόνο για τα τσιγάρα προτείνουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο τυποποίησης, αλλά η πρόθεσή μας εδώ είναι να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει πλήρης ορατότητα και αποτελεσματική απεικόνηση των προεδοποίησεων υγείας. Δεν ε, προβλέπουμε παραδείγματο χάρη μαλακά πακέτα τα οποία είναι, δεν θέλουμε να τα θίξουμε αυτά, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά δεν θέλουμε πακέτα τα οποία μπορούν να είναι ελκυστικά για τους νέους, όπως παραδείγματος χάρη τα πακέτα σε σχήμα κραγιών. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα δούμε και σε λεπτομέρειες και θα τα συζητήσουμε και με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Έχουμε επίγνωση ορισμένων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη σε επίπεδο συσκευασία και πρέπει και αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Προτάθηκε επίσης, η, αναφέρθηκε επίσης ότι οι προδιαγραφές για την συσκευασία θα, έχουν προβλη, θα οδηγήσουν προβλήματα για τη βιομηχανία συσκευασίας που θα έχουν λιγότερη εργασία. Εδώ τονίζουμε ότι ακόμα και αν υπάρξει μια απλοποίηση στη συσκευασία θα υπάρχει πάντα η ανάγκη να παράγονται συσκευασίες και το γεγονός ότι θα είναι θα υπάρχουν εικόνες, θα υπάρχουν ε, προειδοποίηση ασφαλείας, όλα αυτά μπορεί να είναι μια πρόκληση για τη βιομηχανία συσκευασιών και μπορεί να τους δώσει και περισσότερη δουλειά για να συμπεριλάβουν όλα αυτά τα στοιχεία στα νέα πακέτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν και τώρα για να κλείσουμε δίνω το στην εισηγήτρια την ε, Λίντα Μακέβεν. Λίντα, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοντεύουμε πέμπτη απόγευμα και ο κόσμος πρέπει να πάει σπίτι του, οπότε δεν θα σχολιάσω όλα τα λεπτομερή που υπόθηκαν όλες τις λεπτομέρειες. Η κυρία Καρτίνη μίλησε για παραποίηση και για τις ε, προτάσεις και τις εικόνες που υποτίθεται ότι θα οδηγήσουν σε περισσότερη παραποίηση. Δεν υπάρχει όμως καμία ε, απόδειξη για κάτι τέτοιο. Ε, τώρα ήδη το να παραποιήσει κανείς το πακέτο που κυκλοφορεί κοστίζει ίσα ίσα κάποια σέντς, κάποια λεπτά. Το περισσότερο συνδέεται με την τιμή των ε, τσιγάρων παρά με την συσκευασία. Κανένας δεν είπε ότι θα πρέπει να μειώσουμε το, την τιμή των τσιγάρων για να, για να ανταγωνιστούν τα παράνομα που έρχονται από την Λευκορωσία ή οπουδήποτε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τα πραγματικότητα. Η πίεση ασκείται από τη βιομηχανία από όλε τι πλευρέ. Εμεί έχουμε δει, έχουμε εξετάσει το θέμα τη συσκευασία. Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη για το ότι υπάρχει σύνδεση. Η απλή συσκευασία ε, δεν είναι και τόσο απλή, θα έχει φωτογραφίες, ένα σωρό χαρακτηριστικά που μόλι συζητήσαμε. Τα νέα πακέτα θα είναι πολύ πιο ασφαλή λόγω των χαρακτηριστικών ασφαλείας από ό,τι τα πακέτα που κυκλοφορούν τώρα. Η, ε, ε, δεν είναι αλήθεια ότι όταν έχεις μεγαλύτερη εικόνα προειδοποίησης είναι πιο εύκολο να παραποιηθεί. Ε, δεν είναι επιχείρημα που στέκει αυτό. Τα υπόλοιπα ζητήματα ε, νομίζω οι συνάδελφοι έδειξαν έτσι το εύρος απόψεων και την ανάγκη συζήτηση. Εγώ νομίζω πως μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία. Το Συμβούλιο προχωρά πολύ γρήγορα σε συμφωνία στο Συμβούλιο και θέλουν να φτάσουν σε συμφωνία εντός του Κοινοβουλίου και εντός αυτής της Επιτροπής ε, και Οι εισηγητές έχουμε συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, θα αρχίσουμε να συντάσσουμε συμβαστικές, θα λάβουμε υπόψη τα όσα υπόθηκαν εδώ, θα κοιτάξουμε να δεχτούμε τα λογικά αιτήματα, αλλά όχι αυτούς που προσπαθούν να διαγράψουν φυσικά την πρόταση της Κομίσιον, αλλά δεν είναι και η θέση πλειοψηφία της Επιτροπής μας, ούτε και των υπολείπων Επιτροπών. Στις άλλες επιτροπές όντως υπάρχει μια που είναι πιο δύσκολη από ό,τι άλλες, αλλά οι περισσότερες άλλες επιτροπές έχουν προβλήματα με λεπτομέρειες της νομοθεσίας, αλλά όχι με την πραγματική ε, σύλληψη της ίδιας της οδηγίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα βρούμε συμβιβαστικέ και ελπίζω πως οι συνάδελφοι θα έχουν υπόψη τους αυτό που είπατε, Πρόεδρε, για τα νούμερα. 700.000 άνθρωποι το χρόνο. Παρακαλώ αυτό να το θυμάστε και μπορούμε να, κάνουμε, να σημάνουμε τη διαφορά. Και αν όχι, τότε θα πρέπει να το αιτιολογήσουμε στους ψηφοφόρους μας, γιατί οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θέλουν σκληρή δράση, αυστηρή δράση για το κάπνισμα. Θυμάστε πριν λίγα χρόνια όταν μιλήσαμε για απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, ε, θυμάστε τι αντίδραση είχε ένα σωρό κόσμος αντέδρασε. Ναι, στην χώρα μου ε, κανείς δεν το ήθελε εκτός από ένα κόμμα. Ε, γενικά το ευρύτερο κοινό δεν το ήθελε. Κανένας όμως τώρα δεν θέλει να επαναφέρει το κάπνισμα στα εστιατόρια και στα μπαρ. Είχε μεγάλο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία σε όλες μας τις χώρες. Ας είμαστε λοιπόν θαραλέες, είμαστε γενναίοι, ας λάβουμε τις τολμηρές αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε και που έχουμε λάβει και στο παρελθόν και ας μειωθεί ο αριθμός των ε, καπνιστών στο μέλλον. Ευχαριστώ. Έληξε λοιπόν η συζήτηση στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε 10-11 Ιουλίου για το θέμα αυτό. Και προβλέπεται ε, ενδεικτικά για το Σεπτέμβριο στην ε, Ολομέλεια. Τον Ιούλιο, τον Ιούλιο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Ένβη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, όλους τους συμμετέχοντες. Τελευταίο θέμα της ημέρησιας διάταξης, επόμενη συνεδρίαση 19-20 Ιουνίου και να αναφέρω για τους λίγους συναδέλφους ε, που είναι ακόμη εδώ ότι έχουμε ένα workshop για την ασφάλεια των ασθενών από τις 3 και 4 μέχρι τις 6 ASP 1 ε2 θα υπάρχει διερμηνία αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ε, όλοι παρακαλείστε να προσέλθετε, είστε προσκεκλημένοι. Και ε, όλοι όσοι θα επιστρέψουν, ε, καλό μεσημέρι, καλό ταξίδι, ευχαριστώ πολύ.